Małe opóźnienie jest celowe, bo chcemy dać troszkę czasu, aby... Καλησπέρα σας. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε ε, στον Επίτροπο λίγο χρόνο για να συγκεντρωθεί. Γι' αυτό καθυστερούμε λίγο την έναρξη. Σήμερα δεν ήταν εύκολη μέρα. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Χόγκαν θέλω να σας δώσω λίγο χρόνο για να ανασυνταχθείτε. Λοιπόν, δεν ξέρω, θέλετε να κάνετε ε, κάποια σχόλια ή ε, να προσθέσουμε κάτι στην ημερήσια διάταξη ή να συνεχίσουμε λοιπόν με τη συνήθεια διαδικασία. Ε, Έχουμε εδώ τα πρακτικά προς από τη συνεδρίαση της 6ης και 7ης Νοεμβρίου. Εγκρίνονται λοιπόν και μπορούμε να περάσουμε στο βασικό θέμα της απόψινής συνεδρίασης. Να καλωσορίσω τον Επίτροπο κύριο Χόγκαν, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε καιρό που συζητάμε και περιμέναμε να φτάσει 29η Νοεμβρίου Έχουμε ακολουθήσει όλη τη διαδικασία, έχουμε τις διαβουλεύσεις, ακροάσεις, έγγραφα πολλά. Επίσης και προσδοκίες. Πρέπει να σας πω πως από πλευράς ευρωπαϊκού ε, καταναλωτικού κόσμου αλλά και γεωργικού κόσμου οι προσδοκίες είναι μεγάλες. γνωρίζετε κι εσείς μάλλον καλύτερα από ότι εγώ πως η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκε σήμερα το πρωί. Να δούμε ποια είναι τα βήματα τα οποία θα ακολουθήσουν. Δεν θα σας δώσω υπερβολικές λεπτομέρειες. Πάντως μετά την ε, παρουσίαση που θα μας κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσω το λόγο στους συντονιστές. Και μετά ο κύριος Επίτροπος θα απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Και μετά από αυτό θα έχουμε και κάποιο χρόνο στη διάθεσή μας για να ακούσουμε και τα υπόλοιπα μέλη. Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Χωρίς λοιπόν να το καθυστερώ, αγαπητέ συνάδελφοι, θα σας δώσω... Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, θα σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ αξιότιμα μέλη. Είναι χαρά για μένα που είμαι εδώ σήμερα το βράδυ και έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την ανακοίνωση για την ΚΑΠ, την οποία ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νωρίτερα σήμερα. Θα την παρουσιάσουμε και στο Συμβούλιο Γεωργίας όταν θα συνεδριάσει αυτό το Δεκέμβριο. Τώρα, Καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσά έχετε περάσει πολλέ αναθεωρήσει τη ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια, κυρίω το 2013, και ίσω η αντίδραση ήταν Ε, τα έχουμε δει αυτά. Όμως, αυτή, αυτός ο δικός χάρτης για τη μετά το 2020 ΚΑΠ μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια διαδικασία εξελικτική και δεν θα την θεωρούσα επαναστατική. Παρόλα αυτά συμπεριλαμβάνει κάποια πολύ σημαντικά θέματα και αλλαγές που θα βοηθήσουν και την κοινωνία ευρύτερα αλλά και τους ίδιους τους ε, παραγωγούς. Όταν ε, σα συνάντησα για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2014 θα θυμόσαστε ότι μιλήσαμε πολύ για την απλούστευση. Έκτοτε Πέρασαν τρία χρόνια και αυτό μας έδωσε μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή της πολιτικής και πιστεύω πως αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα το πόσο περίπλοκη είναι. Ξέρουμε τι λειτουργεί και έχουμε και μια καλύτερη ιδέα για το τι δεν λειτουργεί. Αυτά τα τρία χρόνια επίσης αντιμετωπίσαμε δύσκολες περιστάσεις σε κάποιες γεωργικές αγορές ε, κυρίως, όχι όμως αποκλειστικά, στα γαλακτοκομικά, στα οποροκυπευτικά ε, και στο χείριου κρέατος. Και καλό είναι να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε πάνω από ένα δις ευρώ σε επιπλέον ε, στήριξη για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις στην αγορά από το Σεπτέμβριο του 2014. Αυτή η χρηματοδότηση είχε πολύ θετικέ επιπτώσει στην αγορά. Είναι όμω σαφέ πω το να κινητοποιήσουμε τέτοιου είδους ποσά στο μέλλον με ad hoc τρόπο δεν είναι βιώσιμη λύση. Χρειαζόμαστε μια διαφορετική απόκριση. Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για το γεωργικό κλάδο και για τους ανθρώπους που εξαρτώνται από αυτόν. Όλοι συμφωνούμε πως η ΚΑΠ ήταν μια μεγάλη επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα είναι το ίδιο σημαντική όσο ήταν το 1962, παρόλο που οι συνθήκες και οι προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή άλλαξαν πάρα πολύ μέσα αυτά τα 50 χρόνια. Η δυνατότητα της πολιτικής αυτής να, αλλάσει, να, να αλλάζει, να προσαρμόζεται, ε, έχουν εξασφαλίσει ότι είναι πετυχημένη και εξακολουθεί να είναι σημαντική. Η σημερινή ανακοίνωση απηχεί μια πολιτική που μεταλλάσσεται για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα. Κάναμε και δημόσια διαβούλευση στην αρχή της χρονιάς 320.000 άνθρωποι στείλανε παρατηρήσεις. Πολύ περισσότερο από την περασμένη φορά που κάνουμε κάποια μεταρρύθμιση που λάβαμε 5.000 περίπου τέτοιου είδους σχόλια. Και η μεγάλη ε, πλειοψηφία των πολιτών και των εμπλεκομένων είναι υπέρ του να ε, πληρώνουμε άμεσες επιδοτήσεις στους παραγωγούς έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των ευρωπαϊκών τροφίμων. Όμως η πλειοψηφία αυτών επίσης πιστεύουν πως η ΚΑΠ θα πρέπει να κάνει παραπάνω για το περιβάλλον και για τις προκλήσεις τη αλλαγής του κλίματος. Η ανακοίνωση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια της προόδου που έχουμε επιτύχει το θέμα της απλούστευση και να δούμε πώς μπορούμε ε, να αντιμετωπίσουμε τους περιορισμούς ε, που αντιμετωπίζουμε, μια και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα βασικά κείμενα. Θέλω λοιπόν να αναγνωρίσω τη δική σας βοήθεια στη διαδικασία της απλούστευσης και να σας πω πως εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας. Από τότε που είναι επίτροπος, έχω ήδη πάντοτε πτονίσει ποιο είναι το τεράστιο δυναμικό του κλάδου ε, των τροφίμων και της γεωργίας και πως υπάρχει μια σειρά από συμπληρωματικές ευρωπαϊκές πολιτικές που είναι πολιτικές ε, προτεραιότητες της Επιτροπής Γιόνκερ. Είναι Μία πολιτική που δεν είναι μόνο σημαντική για τα 7 εκατομμύρια εκμεταλλεύσει οι οποίες λαμβάνουν άμεσες επιδοτήσεις ή για τα 44 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι άμεσα ή έμεσα εξαρτώνται για απασχόληση από τον τομέα των τροφίμων, αλλά και για τα 500 εκατομμύρια καταναλωτές για τους οποίους η ΚΑΠ εξασφαλίζει την ασφάλεια των τροφίμων καθημερινά. Αν το σκεφτούμε αυτό θα δείτε πω η ΚΑΠ έχει έναν ε, άμεσο ρόλο σε σχέση με πολιτικές ε, στην απασχόληση, στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις, στην Ενεργειακή Ένωση και στο δυναμικό αυτής, την κυκλική οικονομία, τη βιοοικονομία, την έρευνα και την καινοτομία που θα φτάσει στις εκμεταλλεύσεις μας, που συνδέει τους γεωργούς και τις κοινότητες στην Ήπεθρο με την ψηφιακή οικονομία και βεβαίως συνεισφέρει στη θεματολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μετανάστευση. Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια στα οποία προσφέρει η Γεωρία και η ΚΑΠ είναι ο κλάδος του ε, περιβάλλοντος και η φιλοδοξία με το κλίμα. Εμείς είμαστε σίγουρα δεσμευμένοι υπέρ της COP21 και μία σύγχρονη ΚΑΠ είναι απαραίτητη για να προσθέσουμε αξία και να έχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας για το περιβάλλον και το κλίμα. Οι επίτροποι Αρίας, Κανιέτε και Βέλα πιστεύουν και οι δύο πως η Γεωργία έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο που καλείται να παίξει. Θα πρέπει η Γεωργία να συνεισφέρει σίγουρα στα, στους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 και αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί. Από το 90. Έχουμε ήδη μία μείωση 24% σε ε, εκπομπές μη ε, ανθρακούχες των αερίων του θερμοκηπίου και πρόσφατες ε, έρευνες δείχνουν πως εξακολουθούν να, να μειώνονται οι εκπομπές αυτές κατά 1,13% κάθε χρόνο. Από τότε που ξεκινήσαμε με το greening, το πρασίνισμα, το 77% της αρρώσιμης γης υπόκειται στις απαιτήσει της ε, άμυψης ποράς και το 14% της αρρώσιμης γης θεωρείται πως είναι ε, η ειδική προστασίας. Επίσης έχουμε τους μόνιμους βοσκότοπους οι οποίοι αποτελούν το 29% της συνολικής γεωρικής ρής και ένα πέμπτο από αυτούς τους ευαίσθητους βοσκοτόπους ορίζεται από πολύ αυστηρούς κανόνες. Λοιπόν, το greening, το πρασίνισμα, ήταν μια περίπλοκη πολιτική και στην εφαρμογή και στη διαχείριση. Έτσι λοιπόν είπαμε πως θα πρέπει το σχήμα το σημερινό να αντικατασταθεί με μια πιο φιλόδοξη και ευέλικτη προσέγγιση που θα έχει μια τριπλή στόχευση σε καλύτερες περιβαλλοντολογικές και κλιματολογικές δράσεις και μεγαλύτερη ε, απλούστευση. Επειδή είναι πολύ διαφορετικές οι εμπειρίες μας στη Γεωργία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν πιστεύουμε πως ένα κουστούμι κάνει για όλους. Είπαμε πως θα πρέπει να κάνουμε μια άλλη ε, επιλογή με εφαρμογή η οποία θα λαμβάνει υπόψη πολύ περισσότερο ε, την επικουρικότητα και θα δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να προτείνουν τα ίδια λύσεις. Άρα λοιπόν δεν θα έχουμε πια τις Βρυξέλλες οι οποίες θα αποφασίζουν ε, πόσο ε, φαρδιά ή στενά θα πρέπει να είναι ε, τα αυλάκια ή πόσα δέντρα θα πρέπει να έχεις σε ένα χωράφι. Όχι, θα αφήνουμε τα κράτη-μέλη να ορίζουν αυτές τις πρακτικές που θεωρούν πως είναι πιο κατάλληλες για τις δικές τους συνθήκες. Και για να μην έχετε αμφιβολίσει ότι αυτό θα προσφέρει στο περιβάλλον, να σας πω πως η νέα όπου η στήριξη Δήματος των γεωργών θα έχει ως ως προϋπόθεση να αναλαμβάνουν κάποιες ε, πρακτικές υπέρ του περιβάλλοντος ε, θα αποτελέσει τη βασική γραμμή για ακόμα πιο φιλόδοξα εθελοντικά σχήματα και καθεστώτα βασικός κόμβος είναι η απλούστευση. Όπως και με το πρασίνισμα, δεν πιστεύουμε πως εδώ πάλι μπορούμε να επιβάλλουμε κάποιες λύσεις ίδιες για όλους. Όχι. Αυτό που προτείνουμε είναι να κάνουμε μια αλλαγή βήμα-βήμα για το πώς η πολιτική μας θα παρουσιάζεται στο μέλλον. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν επιφυλάξεις για αυτή, τη νέα προσέγγιση και σήμερα, μια που είμαι εδώ, θέλω να σας καθησυχάσω. Σας είπα για ποιο λόγο η πολιτική μας ήταν επιτυχή για 50 χρόνια και ένας από τους λόγους είναι το γεγονός πως η ΚΑΠ είναι η κοινή γεωργική πολιτική. Έχουμε μια πολύ πετυχημένη εσωτερική αγορά και έχουμε αποφύγει τις τερβουλώσεις μεταξύ κρατών μελών. Αυτό που προτείνεται εδώ είναι μια σημαντική μετακίνηση στο βάρος ευθυνών και των σχέσεων μεταξύ των τριών βασικών παικτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των κρατών μελών και ε, του παραγωγού, γεωργού ή του ε, ε, γεωργικού κλάδου. Αλλά δεν θα κάψουμε τα χλωρά μαζί με τα ξερά. Όχι σήμερα η ΚΑΠ βασίζεται στη συμμόρφωση με πολύ συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς κανόνες και με ευρύτατους ελέγχους. Στα πλαίσια της περαιτέρω απλούστευσης της ΚΑΠ είναι πολύ περιορισμένο το πεδίο για μεγαλύτερη πρόοδο σύμφωνα με την ε, προσέγγιση βάση συμμόρφωση που ακολουθούμε σήμερα. Αλλά λοιπόν θέλουμε ένα νέο μοντέλο. Περισσότερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή τη πολιτική, λιγότερη γραφειοκρατία για του ε, γεωργού και μια πολιτική που να βασίζεται σε παραδοτέα αποτελέσματα, που θα παρομοιάζει με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αποτελέσματα που στοχεύουν σε καλά, ε, σε ε, θετικούς προπολογισμούς. Άρα λοιπόν θα πρέπει η, να είναι πιο φιλική προς το χρέος, πιο απλή και πιο σύγχρονη η πολιτική μας, έτσι ώστε οι προκλήσεις να μετατραπούν σε ευκαιρίες. Έτσι λοιπόν θα περάσουμε από τη συμμόρφωση στα παραδοτέα αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν τότε να εντοπίσουμε ξεκάθαρα ποιοι είναι οι στόχοι μα που θα πρέπει να πετύχουμε και σε ποιο επίπεδο. Καταρχήν, οι στόχοι αυτοί θα τεθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει κάθε ε, κράτο μέλο ή περιφέρεια να σχεδιάσει ένα στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ. Δηλαδή, τι σημαίνει μία εκ των προτέρων αξιολόγηση να εντοπίσουν τι ανάγκε του και μετά να ορίσουν του στόχου και τον τύπο των δράσεων που θα του βοηθήσουν να πετύχουν του στόχου αυτού. Που θα είναι ε, προσδιορισμένο στη βασική πράξη και θα έχουμε αποσυνδεδεμένη ε, στήριξη, συνδεδεμένη στήριξη, επενδυτική στήριξη και περιμοντολογικέ δράσει. Το σχέδιο τη ΚΑΠ υπόκειται σε έγκριση σε κάθε περίπτωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα εξετάζει τη στρατηγική που προτείνεται βάσει στα τεκμήρια που θα προσκομιστούν και θα πρέπει να υπάρχει συνοχή με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους στόχους των κρατών μελών και βέβαια να είναι ε, σε απόλυτη συνοχή με ε, τους στόχους και τους ε, χρηματοδοτικούς φακέλους που επιλέγουν τα κράτη-μέλη. Αυτή η προσέγγιση σημαίνει πως θα έχουμε στόχους και μέτρηση απόδοσης σε επίπεδο κράτους μέλους. Η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του παραγωγού θα απλουστευτεί σε μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε το κράτος μέλος θα επιβάλλει τις υποχρεωτικές δεσμεύσεις στο επίπεδο της εκμετάλλευσης. Ένα ακόμα σημείο στο οποίο μπορούμε να μειώσουμε το ε, πόσο περίπλοκοι είναι, είναι οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμμόρφωση που θέλει να πετύχει συγκεκριμένες ε, συγκεκριμένα αποτελέσματα. Είναι πολύ περίπλοκα και θα πρέπει να τα ορίσουν τα κράτη-μέλη. Αυτή λοιπόν η πιο ελαφριά προσέγγιση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μπορεί να οδηγήσει, και αυτή είναι μια επιφυλαξή, τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν μη ε, απαραίτητες υποχρεώσεις στους δικαιούχους. Στα πλαίσια τη εξέταση των σχεδίων για την ΚΑΠ το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, προσπαθήσει να εξετάσει προσεκτικά έτσι ώστε να μην έχουμε νομοθετικό υπερθεματισμό. Η γραφειοκρατία στο επίπεδο του δικαιούχου θα μειωθεί και θα χρησιμοποιήσουμε τη μοντέρνα τεχνολογία, την τεχνολογία τη δορυφορική, την, την ε, υψηλή τεχνολογία έτσι ώστε να μην έχουμε τήσει σε χαρτί και φυσικούς ελέγχους. Ελπίζω ότι έτσι σας ε, ότι παρόλο που έχουμε αυτή την αλλαγή θα παραμείνει κοινή η κοινή γεωργική πολιτική. Και θα ήθελα να μιλήσω και για κάποια άλλα κομμάτια της ανακοίνωσης. Είμαι απολύτως ε, ε με τα προβλήματα που έχουν οι νέοι γεωργοί. Γνωρίζουμε ότι μόνο το 6% των γεωργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτω από 30 ετών, ενώ το 50% είναι από 55 και πάνω. Να σας θυμίσω ότι στη μεταρρύθμιση του 2013 η πληρωμή για τους νέους γεωργούς ήταν η ανώτατη κάλυψη των άμεσων πληρωμών. Συνολικά χρηματοδοτήσαμε πέρυσι περίπου 280.000 γεωργούς με κόστος 3 δις και 177.000 νέοι γεωργοί προγραμματίζεται να λάβουν στήριξη στα πλαίσια της ανάπτυξης της υπαίθρου. Η ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου λέγει ότι η στήριξη άμεσων πληρωμών δεν βασίζεται σε υγιείς εκτιμήσεις και ε, δεν δίδεται πάντα στους νέους γεωργούς οι οποίοι την έχουν ανάγκη. Δεν υπάρχει σωστή σωστό συντονισμός ανάμεσα στις πληρωμές και στους δύο πυλώνες και ακριβώς για αυτούς τους λόγους το θέμα της ενθάρρυνσης, της γενεακής ανανέωσης πρέπει να ειδωθεί σαν συνεργατική προσπάθεια ανάμεσα στην Ένωση και τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέσα όπως η φορολογία, το κληρονομικό δίκαιο και οι χωροτακτικές ρυθμίσεις. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την συνεκτικότητα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές δράσεις. Νομίζω ότι έτσι θα καλύψουμε καλύτερα τις ανάγκες των νέων γεωργών. Ένα επιπλέον σημείο είναι το θέμα της ε, επιφανειακής ανισότητας ή ε, αδικίας αν θέλετε στην κατανομή των πληρωμών ανάμεσα στους γεωργούς. 80 με 20 υποτίθεται είναι ο λόγος, η σχέση στις πληρωμές, όπου το 20% των γεωργών παίρνουν το 80% των πληρωμών. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν παραδεχτούμε τη συγκεκριμένη αυτή, τον συγκεκριμένο ισχυρισμό ότι καλύπτουμε το σύνολο της ε, περιγραφής της κατάστασης. Ότι δηλαδή το 72% της άμεσης βοήθειας πληρώνεται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ανάμεσα σε 5 και 250 εκτάρια που είναι οικογενειακού τύπου. Το θέμα της δικαιοσύνης στην κατανομή των πληρωμών είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιδιωχθεί περαιτέρω και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως και στο παρελθόν. ανώτατο ύψος, αν θέλετε, των άμεσων πληρωμών, μειούμενες πληρωμές ε, στα πλαίσια της μείωσης της στήριξης για μεγάλες γεωργικέ εκμεταλλεύσεις και αναδιανεμητικές πληρωμές έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε με στοχευμένο τρόπο τις μικρομεσές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Και φυσικά βοήθεια στους πραγματικούς, τους γνήσιους γεωργούς. Βέβαια η τελευταία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, για υποχρεωτικά ανώτατα όρια απερίφθη από τους συνομοθέτες, οπότε θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Εν πρέπει να δούμε ότι για τις ε, διεκδικήσεις εισαγωγικά του 2016 εννέα κράτη-μέλη ε, θα εξαντλήσουν τις πληρωμές και ένα δέκατο θα το κάνει το 17. Σε σχέση λοιπόν με θέματα δικαιοσύνης, η κοινή αγροτική πολιτική πρέπει να παίξει τον ρόλο της, τον πραγματικά προσπαθώντας να εξισορροπήσει τις αρχές της ισότητας ανάμεσα στα κράτη-μέλη, μικρά ή μεγάλα, ανατολικά ή δυτικά, βόρεια ή νότια. Αυτό το υπενθύμησε και ο πρόεδρος Ιούνκερ. Ακόμα και αν η διαφορετικότητα στο κόστος της εργασίας, στο κόστος της γης και οι διαφορετικές αγρονομικές δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ληφθούν υπόψη, οι προκλήσεις είναι θα έλεγα αντίστοιχες για όλους τους γεωργούς. Θέλω να συμπληρώσω και κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Η ανακοίνωση καλύπτει πολλούς τομείς στους οποίους η κοινή αγροτική πολιτική μπορεί να ενισχύσει τις περιοχές της υπαίθρου, δημιουργώντας θέσεις εργασίας ιδιαίτερα στην αναδυόμενη βιοοικονομία που έχει τεράστιο δυναμικό για την αναγέννηση αν θέλετε ε, την δημογραφική των περιοχών αυτών. Ξέρω ότι κάποιοι από εσά ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το λεγόμενο FES χωριό, το Smart Village, την πρωτοβουλία αυτή. Και χαίρομαι που η ανακοίνωσή σας αναγνωρίζει την προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας ευχαριστώ για την στήριξή σας όπως και την στήριξη της Επιτρόπου Κρέτου. Ο ρόλος επίσης της ψηφιακής προόδου στις αγροτικές περιοχές είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Η μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας στις περιοχές της υπαίθρου. Ε, οι ανάγκες και οι συνεισφορές των γεωργικών περιοχών θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται και στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της μελλοντικής κοινή αγροτικής πολιτικής. Αυτό είναι κάτι που ο Επίτροπος Μοέντας και εγώ ε, ζητούμε από κοινό. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι όλοι οι γεωργοί έχουν πρόσβαση σε ένα σύστημα παροχής σύμβουλων όπου εκπαιδευμένοι σύμβουλοι, ε, ενημερωμένοι μπορούν να δώσουν την τεχνολογία και τις μεθόδους παραγωγής της φιλικές για το περιβάλλον που χρειάζονται οι παραγωγοί και σε σχέση με την βιώσιμη γεωργική παραγωγή και στον τομέα της υγείας, της διατροφής, των αποβλήτων τροφίμων και της ευημερία των ζώων. Μπορεί να κάνει σε όλους αυτούς τους τομείς περισσότερα εκείνη η αγροτική πολιτική και σε σχέση, δίνω ένα παράδειγμα, με την αντιμικροβιακή αντοχή όπως ε, περιγράφεται στην πρωτοβουλία One Health. Έτσι λοιπόν μπορούμε να βοηθήσουμε επίσης και στην προώθηση υγιέστερης διατροφής, να βοηθήσουμε το πρόβλημα της παχυσαρκίας, της κακής διατροφής και αυτό είναι κάτι το οποίο επιδιώκουμε μαζί με τον Επίτροπο Άντριου Καΐτης. Θέλω να θυμίσω επίσης πως εμείς προσπαθούμε να ακολουθήσουμε και τους προσανατολισμούς της αγοράς. Η σημερινή ανακοίνωση είναι αυτή που θα μας κατευθύνει τα επόμενα χρόνια στον ίδιο δρόμο που ακολουθούσαμε μέχρι τώρα. Υπάρχουν πολλά τα οποία θα μπορούσα να πω περισσότερα, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε κάποιο χρόνο για να περάσουμε σε λεπτομέρειες. Εύχομαι να λάβετε υπόψη την ανακοίνωση αυτή, η οποία νομίζω ότι είναι μια σημαντική συνεισφορά για την προετοιμασία της νομικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το επόμενο έτος. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και να περάσουμε στην συζήτηση, ερωτήσεις. Παρακαλώ πολύ προσέξτε το χρόνο. Κοιτάξτε, έχετε δύο λεπτά. Θα δώσω το λόγο καταρχήν στους συντονιστές. Δύο λεπτά για τον κάθε συντονιστή. Ο κύριος Τέσ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε και θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά την κατάσταση στην κοινή αγροτική πολιτική δεν πρόκειται για επανάσταση αλλά χρειάζονται διορθώσεις στους τομείς αυτούς όπου είναι απαραίτητο αυτό. Είναι πολύ λογικές οι προτάσεις σας. Εμείς θα τις συμπληρώσουμε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλουμε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν τομείς ε, στους οποίους θα πρέπει να δουλέψουμε για να κάνουμε και τις δικές μας προτάσεις. Βεβαίω, η αγροτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τι σοβαρότερε συνιστώσει της Ένωσης. Και εδώ και πολλά χρόνια παρακολουθώ αυτό το θέμα της αγροτικής πολιτικής, παρακολουθώ τη δραστηριότητα των Ευρωπαίων ε, αγροτών. Εκεί που λίγο έχω επιφυλάξεις είναι με το θέμα των πολλών εθνικών αρμοδιοτήτων που ενισχύονται. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να είμαστε προσεκτικοί εκεί που είναι θέματα εθνικής αρμοδιότητας να μην υπάρχει στρέβλωση ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η κοινή αγροτική πολιτική να παραμείνει ευρωπαϊκή πολιτική. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι τα κονδύλια τα οποία δαπανώνται για τους γεωργούς και τα οποία δεν ε, ε, απορροφούνται πάνε 40% συγκεκριμένα στις ε, αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Θα πρέπει κάθε φορά λοιπόν να εξηγούμε, να είναι στη δημόσια συζήτηση για ποιο λόγο υπάρχουν εκατομμύρια τα οποία είναι προς διάθεση στους ε, γεωργούς και να πηγαίνουν στους πραγματικούς δικαιούχους, να πηγαίνουν σε προγράμματα τα οποία πραγματικά πρέπει να χρηματοδοτούν όπως αρχικά είχαμε βλέψει. Και αυτό θα πρέπει να γίνει με μεγάλες διευκρινήσεις πριν το τέλος της δικής μας θητείας. Πρόεδρος, θέλω να σας πω ότι έχουμε τον κύριο Σιπ Χούμπερ που ήταν παλαιό μέλος και είναι σήμερα επισκέπτης εδώ. Θα ήθελα να σας ευχηθούμε κάθε καλό και ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Επίσης, έχουμε τον κύριο Αχτουή, πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Καλώς ορίσατε και θα δώσω το λόγο στον κύριο Άντριο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ε, παρουσίασή σας. Βεβαίως θα επανέλθουμε στην ε, δηλωσή σας και θα την επεξεργαστούμε. Μιλήσατε για την ε, αυλοποίηση. Εγώ συμφωνώ με αυτό που παρουσιάσατε, ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στην γενικότερη μεταρρύθμιση, να μην επανέλθουμε σε πολλές επανεθνικοποίησεις. Αν κατάλαβα καλά αυτό που μας είπατε, λέτε ότι πρέπει να υπάρχει ένα κοινό ε, θεμέλιο και όσον αφορά την επικουρικότητα να αφιερώσουμε στην υλοποίηση κάποια μέτρα που να είναι μέτρα που απορρέουν από αυτήν την πολιτική. Μιλήσατε επίσης για το κλίμα, μιλήσατε για το περιβάλλον. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ανσωματώνεται αυτές τις πτυχές. Η γεωργία είναι στην καρδιά της ε, κοινωνίας και μιλάτε επίσης πολύ για την απασχόληση. Χαίρομαι γιατί εμείς εδώ έχουμε κάνει πολλή δουλειά για το θέμα της απασχόλησης. Το ενσωματώνεται στη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Επίσης, να μιλήσουμε και για την αγορά δεν αλλάζει τίποτα. Εδώ θα είμαι λιγότερο ενθαρρυντικός και θετικός. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τις διακυμάνσεις. Αυτά που μας παρουσιάζεται εδώ σίγουρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν απαντήσεις σε κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στο μέλλον. Το θέμα της ρύθμισης. Εδώ θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα αυτό με άλλα εργαλεία από αυτά που μας προτείνεται. Υπάρχουν νέοι γεωργοί τους οποίους στοχεύεται με συγκεκριμένα μέτρα. Παραδείγματο χάρη για την εγκατάσταση των νέων γεωργών, των νέων αγροτών. Εδώ πραγματικά θα πρέπει να δούμε αν αυτά τα μέτρα αρκούν ή αν χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Σίγουρα λοιπόν, και αυτή είναι μια γενική παρατήρηση, χρειάζεται συνοχή Όσον αφορά την γενικότερη, αν θέλετε, πολιτική σας, θα πρέπει να δούμε τα θέματα κοινωνία. θα πρέπει να θέλουμε τα θέματα της γεωργίας και να δούμε τι επιπλέον θα πρέπει να προσθεθεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν να πω ότι χαιρετίζουμε τη δήλωση του Επιτρόπου, σαφώς και Πολλά από τα σημεία που είχαμε υποβάλει έχουν συμπεριληφθεί. Είναι πολύ σημαντικό από πού ξεκινήσατε και πού καταλήξατε, κύριε Επίτροπε. Θυμάμαι την τελευταία συζήτηση για την δημιουργία της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Το θέμα του προϋπολογισμού όμως κύριε Επίτροπε, όπως όλοι ξέρουμε με το Brexit θα υπάρξουν συνέπειες στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Και βεβαίως η συζήτηση και η διαπραγμάτευση για το Brexit σίγουρα θα μας βοηθήσει να μειώσουμε την ε, μαύρη τρύπα που θα προκύψει από το, την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει πίεση στον προϋπολογισμό και βεβαίως το θέμα της επέμβασης των Βρυξελών στην πολιτική είναι κάτι που πρέπει να το δούμε προσοχή. Το θέμα δεν είναι ε, οι Βρυξέλλες και κατά πόσο παρεμβαίνουν. Το θέμα είναι πώς ερμηνεύουν ε, οι εθνικές αρχές και πώς υλοποιούν τους κανονισμούς των Βρυξελών. Χρειάζεται η κατεύθυνση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στα τρόφιμα και στη γεωργία και μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να υπάρξει συνοχή. Είπατε πολύ σωστά την συνεισφορά της γεωργίας για θέματα περιβάλλοντος και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Βεβαίως θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες όσο προχωράμε και θα συμφωνήσω με τον Άλμπερντες όταν έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία για τον προϋπολογισμό και τις γεωργικές δαπάνες. Σας ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις σας. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε μέσα στο χρονικό διάστημα που έχουμε να φτάσουμε σε μία συμφωνία και ελπίζω ότι και οι δικές μας προτάσεις από εδώ και πέρα συμπληρωματικές θα ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για τις δηλώσεις σας. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, καταλαβαίνω ότι θέτετε ένα πλαίσιο, στόχους, μιλάτε για απλοποίηση, μιλάτε για συναπόφαση. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Λέτε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος περιθώριο ελιγμού για τα κράτη-μέλη. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Ε, σκέφτομαι εδώ τη δική μου χώρα, και έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα είναι πολύ περίπλοκα. Πώς ε, θα προχωρήσουμε με μια κοινή αγροτική πολιτική. Υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα και πολλές δυσκολίες. Και με απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της τρέβλωσης του ανταγωνισμού. Γιατί υπάρχουν χώρες με πάρα πολύ αυστηρούς περιβαλλοντολογικούς κανόνες, κανόνες για την προστασία και την ευημερία των ζώων και άλλα κράτη χωρίς. Αυτό σαφώς και δημιουργεί τελείως διαφορετικά μέτρα και σταθμά και στρέβλωση ανταγωνισμού. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Όλοι θέλουμε να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της γεωργίας, αλλά θέλουμε η στήριξη να πηγαίνει σε πραγματικούς αγρότες. Και εδώ έχουμε παραδείγματο χάρη ε, κτηνο, τοφικές μονάδες, με 40 αγελάδες, με κάποιες διαφορετικές δραστηριότητες οι οποίες συνεχίζουν να παίρνουν επιδόματα τα οποία δεν αντιστοιχούν στην δραστηριότητά τους. Κοιτάξτε, στην Γερμανία πολύ πρόσφατα είδαμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τα σφαγεία, με τη μεταφορά των ζώων. Είδαμε σε μία εκπομπή πολύ πρόσφατα στη γερμανική τηλεόραση να μεταφέρονται ζωντανά ζώα με άθλιες συνθήκες. Είναι δυνατόν αυτά να συμβαίνουν στην Ευρώπη, μέσα στην Ευρώπη. Είναι δυνατόν στην Ευρώπη να μην μπορούμε να εφαρμόσουμε και να τηρήσουμε τα ελάχιστα αυτά προαπαιτούμενα για τη μεταφορά των ζώων. Δεν είναι δυνατόν να μεταφέρονται τα ζώα προσφαγή σε τρίτες χώρες ή από τρίτες χώρες με αυτές τις άθλιες συνθήκες. Κύριε Επίτροπε, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα, θέματα που αφορούν και τους γεωργούς και το περιβάλλον και οι μεγάλες μεταφορικές εταιρείες δεν μπορεί εδώ να παραβιάζουν καθημερινά την ευημερία των ζώων. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χόγκαν, μας παρουσιάσατε εδώ την ΚΑΠ ως επιτυχία. Εξηγήστε με λοιπόν, πού την είδατε την επιτυχία, για ποιον και πότε. Γιατί από το 2003 μέχρι το 2013 εξαφανίστηκε ένα τρίτο των μικρών εκμεταλλεύσεων, γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μου μοιάζει τόσο πετυχημένο αυξάνεται η ηλικία του γεωργικού πληθυσμού. Γερνάει. Είναι ένα θέμα που συζητάμε συνέχεια. Δεν υπάρχει επόμενη γενιά για να αναλάβει. Εγκαταλείπουν την ύπεθρο φέτος και δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώσουμε ε, τι επιπτώσει έχει αυτό σε κάποιες χώρες, σε περιοχές όπως η Γαλλικία, ε, στην Πορτογαλία ή οι δασικέ πυρκαγιέ που έχουν να κάνουν με την εγκατάλειψη αυτών των γεών και όλα αυτά είναι τα αποτελέσματα τη ΚΑΠ κρίσεις, χαμηλές τιμές, δυσκολίες για τους παραγωγούς για να επιβιώσουν κάθε χρόνο. Οπότε, εγώ νομίζω κύριε Χόγκαν πως όλα αυτά δεν είναι μάνα εξ ουρανού και δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη ξαφνικά. Είναι οι επιπτώσεις της ΚΑΠ. Αυτό πρέπει να εξηγήσουμε. Γιατί καταλήξαμε σε αυτές τις συνέπειες μέσω της ΚΑΠ. Και εσείς εξακολουθείτε να προσπαθείτε ε, να ε, υπονοείται πως η Ευρώπη πρέπει να τρέφει τον υπόλοιπο κόσμο και λέγεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ε, γεωργικών ε, διατροφικών προϊόντων. Ελεύθερο εμπόριο, μεγαλύτερη συμμετοχή στις αλυσίδες που θα επέτρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τις εξαγωγές για να ανταποκριθεί στα όσα ζητάει η μεσαία τάξη σε όλο τον κόσμο. Πού είναι η αλληλεγγύη, πού είναι ο χώρος για το γεωργικό πληθυσμό, έτσι ώστε και οι αγρότες των χωρών που ε, αναπτύσσονται να παράγουν οι ίδιοι για τη δική τους μισέα τάξη τα προϊόντα που χρειάζονται. ε, ξέρετε που περιγράφετε τις πολιτικές μας και ξέρετε που οδήγησαν στη Μεσόγειο. Και τι γίνεται με τον αγροτικό κόσμο, την αγροτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο περισσότερες εξαγωγές, τόσο λιγότερο εισόδημα. Και το ξέρετε. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τι θα κάνετε τι θα κάνετε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε δίκαιες τιμές. Και επειδή βλέπω τον πρόεδρο με το σφυρί στο χέρι, θα κλείσω λέγοντας πως δεν έχω λόγια ε, που χρειάζονται. Τι έγινε, τελείωσε ο χρόνος μου. Ε, λοιπόν, ψάχνω λέξεις κλειδιά στην ανακοίνωσή σας. Δίκαιες τιμές, ρύθμιση της παραγωγής, γεωργική οικολογία, ε, ευζοία των ζώων και το κλίμα στην, ε, στον πυρήνα μιας δημόσιας και υγιούς γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω να σας πω το εξή. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Γιατί ε, θα νομίζετε ότι το κάνω προσωπικά προς εσάς. Ο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, σήμερα η τίτλη στον τύπο ήταν ότι θέλετε να καταργήσετε το πρασίνισμα και ότι επανεθνικοποιείτε η κοινή αγροτική πολιτική. Αυτή είναι η καρδιά της μεταρρύθμισής σας. Με την επανεθνικοποίηση λέτε ότι καταργείτε τη γραφειοκρατία. Μα τα εθνικά κράτη είναι αυτά που έκαναν ακόμα πιο περίπλοκα τα πράγματα στην τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Θα ήθελα να ξέρω αν τελικά έχουμε 28 διαφορετικές εφαρμογές και υλοποιήσεις αυτής της νέας μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Μα τα πράγματα θα είναι ε, τελικά εντελώς διαφορετικά από το ένα κράτος στο άλλο. Ας παραμείνουμε λοιπόν Ευρωπαίοι, ας παραμείνει ευρωπαϊκή η κοινή αγροτική πολιτική. Θέσατε κάποιους στόχους. Αναφερθήκατε στο περιβάλλον ε, ακροθυγός και η τελευταία μεταρρύθμιση είχατε πολύ συγκεκριμένους στόχους για τη βιοποικιλότητα. Εδώ δεν αναφέρατε τίποτα τέτοιο. Λέτε ότι πρέπει η γεωργία να είναι φιλική προς τις ε, αλλαγές του κλίματος. Κάτι πρέπει να αλλάξετε τότε, γιατί δεν βλέπω τίποτα τέτοιο. Κάπως αναφέρατε και την ψηφιακή ε, τεχνολογία. Ναι, σήμερα μιλάμε για την ψηφιοποίηση σε όλους τους τομείς και κατά κάποιο τρόπο είναι το σύγχρονο μήνυμα αν θέλετε. Σε όλους τους τομείς προσθέτουμε ψηφιοποίηση για να δείξουμε ότι κοιτάμε προς το μέλλον. Αλλά νομίζω ότι μιλάτε και για καλύτερη κατανομή στις μεγάλες, στις μικρές επιχειρήσεις. Ούτε εδώ δεν βλέπουμε τίποτα. Πραγματικά κάτι λείπει. Κάτι λείπει κύριε Επίτροπε. Συγκεκριμένες προτάσεις και στόχοι. Συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες πραγματικά λείπουν από αυτό το μικρό έγγραφο το οποίο μας παρουσιάζεται. σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσούλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν διάβασα τον τίτλο της ανακοίνωσής σας, το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας, Κατά κάποιο τρόπο είδα ότι μπορεί να δει κανείς αυτές τις δύο λέξεις μαζί επιτέλους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη τις σοβαρές προτάσεις που γίνονται για τον μετασχηματισμό της κοινή αγροτικής πολιτικής σε μια κοινή αγροτική και πολιτική τροφίμων. Όταν όμως διάβασα το περιεχόμενο για τη διατροφή δεν βρήκα τίποτα, μα τίποτα. Να σας υπενθυμίσω ότι επανειλημμένα το είχα πει όπως και άλλοι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μια ουσιαστική διαφθρωμένη στρατηγική στον τομέα της παραγωγής τροφίμων που θα της επέτρεπε να μην εξαρτάται από τρίτες χώρες για να καλύπτει τις ανάγκες της σε τρόφιμα. Μια στρατηγική που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, πώς να αυξήσουμε την παραγωγικότητα χωρίς να επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Αυτή τη στρατηγική δεν την έχουμε και από ό,τι διαβάζω δεν θα την έχουμε κιόλα. Ο δρόμος τον οποίο ακολουθείτε εσείς είναι ας δούμε τι θέλουν οι καταναλωτές και ας καλύψουμε τις ανάγκες τους. Μα μπορεί μια τέτοια λογική να αντιμετωπίσει το θέμα της παχυσαρκίας ή πραγματικά της παρασκευής από τις πολυεθνικές ε, κακού τύπου τροφίμων. Έχουμε ανάγκη από μια στρατηγική η οποία θα πρέπει να προσανατολίσει διαφορετικά τους πολίτες και να στηρίξει τη γεωργία ως προς την παραγωγή τροφίμων. Αν δεν έχουμε μια τέτοια στρατηγική φοβάμαι ότι θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα εξυπηρετεί αυστηρά τα μεγάλα εμπορικά συμφέροντα. Έχετε μια μεγάλη ευκαιρία λοιπόν, σας ζητώ να μην την χάσετε Θέλετε μια πραγματική πολιτική για τους πολίτες ή για τις πολυεθνικές μήπως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πραγματικά αυτά που ακούω από κάποιους όπως τον κύριο Ντες πραγματικά με εκπλήσουν. Πραγματικά τι λέτε όσον αφορά τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Αυτό είναι πραγματική προδοσία. Στη τελευταία μεταρρύθμιση, την οποία θεωρείται επιτυχή, έχουμε 700 αυτοκτονίες το χρόνο. Αυτά είναι τα νούμερα. Αυτή είναι η επιτυχία. Μας παρουσιάζεται μια κοινή αγροτική πολιτική που εξάγει περισσότερο, πιο πράσινη, πιο φιλική προς το περιβάλλον. Πρόκειται για μια γενική παρουσία, η οποία βεβαίως εδώ μας κρύβει ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των παλιών και των καινούριων κρατών μελών και κάποιων ε, σημαντικών διαφορών μεταξύ των διαφορετικών γεωργικών συστημάτων. Και την ίδια ώρα είναι αδύνατον να μην λαμβάνουμε υπόψη μας σήμερα τα οικονομικά βάρη των αγροτών. Διαπραγματεύεστε μια συμφωνία με τις χώρες του Μεκροσούρ και Παραδείγματο χάρη υπάρχουν προϊόντα από τη Βραζιλία που απαγορεύεται να εισάγονται, περνάνε μέσα από τη Ρωσία. Θα πρέπει να σταματήσετε να διαπραγματεύεστε συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου γιατί η οικονομία σας εξαρτάται πάρα πολύ από τις αγωγές και τις εξαγωγές. Εδώ και δεκαετίες η πολιτική σας η οποία οδηγεί στην υπερσυγκέντρωση, στην εξαφάνιση των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, καταργεί και καταστρέφει, τουλάχιστον στη Γαλλία, χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Και επίσης συνδέεται και την πολιτική σας με την πολιτική της μετανάστευσης. Διαθέλετε να εγκαταστήσετε μετανάστες στην ύπεθρο και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Όπως σας είπα και προηγουμένως, θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο. Θα του ζητήσω να απαντήσει στις μέχρι τώρα ερωτήσεις και κατόπιν θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπο, έχετε το λόγο. Να πω επίσης ότι έχουμε και αρκετούς άλλους προσκεκλημένους σήμερα προσκεκλημένους του κυρίου Τεκάστρο και της κυρίας Μαγκίνες. Τους καλωσορίζουμε και αυτούς. Συμμετέχετε σε μια συνεδρίαση που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική και ελπίζω ενδιαφέρουσα. Καλώς ήρθατε όλοι λοιπόν και δίνω το λόγο πάλι στον Επίτροπο Χόγκαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. αναφέρθηκε στον νέο τρόπο, αν θέλετε, λειτουργίας του συστήματος, όπως επίσης και στις δικές μου παρατηρήσεις ξεκαθάρισα τις προθέσεις μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσουν για τους στόχους, όπως το κάνουμε σήμερα σε σχέση με την κοινή αγροτική πολιτική, ζητάμε από τα κράτη-μέλη να καταθέσουν προτάσεις για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς θα βάλουμε στόχους και στην παροχή των διευκολύνσεων και θα προσμετρήσουμε επίσης τις επιδόσεις μας. Η χρηματοδοτική διαθήρηση ε, την οποία έχουμε σήμερα θα συνεχιστεί. Τα μέτρα για την αγορά και όλα τα μέσα τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα και το 2015 και το 2016 για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν ορισμένα προϊόντα θα συνεχίσουν. Το ότι δεν αναφέρθηκα σε αυτά δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζονται. Και συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε για τη σημασία της διατήρησης της κοινή αγροτικής πολιτικής είναι κάτι το, το οποίο με βρίσκει σύμφωνο. Ε, δεν θα υπάρξουν λοιπόν εφόσον μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά μέτρα στρέβλωσης του ανταγωνισμού και θα υπάρξει προστασία της εσωτερικής αγοράς. Αναφερθήκατε και στη διαχείριση των κινδύνων έτσι ώστε να καταφέρουν να διασχίσουν τις ε, περιόδους κινδύνου. Η Γεωργία αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τη σειρά προτάσεων Omnibus σχετικά με το μέσο σταθεροποίησης του εισοδήματος, με την επιπλέον στήριξη των παραγωγών στα πλαίσια των ρυθμίσεων για τον ανταγωνισμό. Όλα αυτά είναι παραδείγματα στα οποία μπορούμε να επενδύσουμε και θέλουμε μέσα από τις προτάσεις μας να βοηθήσουμε τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν τις διακυμάνσεις των τιμών, να, αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της ξηρασίας, των σεισμών, τις πλημμύρες που είδαμε και συναντήσαμε το 16 και το 17, τα θέματα αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν και απαιτούν συγκεκριμένους οικονομικούς πόρους αλλά και νομοθετικά μέσα για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να τα αντιμετωπίσουν. Και είπα ότι η πολιτική διαχείριση της υπαίθρου ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική στις χώρες που αντιμετώπισαν φυσικές καταστροφές και η βοήθεια την οποία δώσαμε και για τους γεωργούς και τους άλλους κατοίκους των περιοχών της Υπέθρου είναι κάτι το οποίο οδήγησε τα κράτη-μέλη να εκφράσουν την ικανοποίησή τους για την παρέμβασή μας. Άλλοι ομιλητές αναφέρθηκαν σε κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις, ε, κ. Νίκολσον συγκεκριμένα. Τώρα το που θα καταλήξουμε αυτό θα εξαρτηθεί από τους συνομοθέτες. Εμείς θα κάνουμε τις προτάσεις μας, και θα δούμε από εκεί και πέρα με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να δεχθούμε τις προτάσεις αυτές. Σας επενδύσουμε λοιπόν ιδίω το Omnibus. Είναι ένα καλό παράδειγμα σχετικά με την υιοθέτηση μέτρων με μεγάλη ταχύτητα, πολιτική βούληση και σωστή κατάληξη. Τα σενάρια για τον προϋπολογισμό είναι δύσκολα και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί σε σχέση με ε, τις επόμενες προτάσεις για το επόμενο, με τις προτάσεις για, το επόμενο νέο για την επόμενη νέα δημοσιονομική περίοδο. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά λόμπι, ιδιαίτερα στους υπουργούς οικονομικών η εφαρμογή των πολιτικών αυτών και χρονοδιαγράμματα για τις πολιτικές αυτές. Νομίζω ότι κάποιες πρώτες προτάσεις θα υπάρξουν τον Ιούνιο και εφόσον το πετύχουμε θα καταφέρουμε νομίζω να ολοκληρώσουμε την πρόταση πριν από τις ευρωεκλογέ. Αυτή είναι και η επιθυμία σας. Νομίζω λοιπόν ότι θα είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε την εφαρμογή των προτάσεων μας όχι μια επαναστατική πολιτική όπως το 2013, αλλά μια εξελικτική πολιτική, σταδιακή ε, και αυτό θα το πετύχουμε το ταχύτερο δυνατόν αυτή τη στιγμή γίνει δεκτή η νομοθετική πρόταση. Αναφερθήκατε και στην ευημερία των ζώων. Στην ανακοίνωση αναφέρεται η ευημερία των ζώων επτά φορές. Είναι κάτι το οποίο θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό δεν ξέρω για κάποια προγράμματα της τηλεόρασης, είναι λανθασμένα αν πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τίποτα για τα θέματα αυτά. Ίσα ίσα χρησιμοποιούμε και αρκετά χρήματα στα πλαίσια της ανάπτυξης της υπαίθρου για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν θέματα ευημερία ζώων. Είναι θέμα του κυρίου Αντρουκάητης περισσότερο, αλλά θα ήθελα να το διευκρινίσω. Τώρα, οι διαφορές και οι οι αλλαγές των διαφορών είναι δεδομένες. Ε, η λογική του one size fits all, ε, ένα μέτρο και το ίδιο για όλους, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει δεκτό. Και αυτό μας δίνει την δυνατότητα να συλλέξουμε τοπικές προτάσεις, οι οποίες καλύπτουν και τους στόχους της Ένωσης. Οι, στη οι γεωργοί στη Φιλανδία έχουν διαφορετικές ανάγκες από τους γεωργούς στην Ελλάδα σε συγκεκριμένους τομείς πρέπει λοιπόν να διαχειριστούμε τη διαφορετικότητα η οποία υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν μόνο μέσω της ευελιξίας να ρυθμιστούν όλα, αλλά είναι και αυτό ένα μέσο. Ε, θα πρέπει επίσης να ενισχύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται ε, πραγματικά με τη γη και καλλιεργούν τη γη, ακόμα και η ε, μερικής απασχόλησης γεωργή. Υπάρχουν μερικοί απασχόλησης γεωργοί και του καλύπτουμε και αυτού και το κάνουν διότι προφανώ δεν του καλύπτει οικονομικά η πλήρη αγροτική δραστηριότητα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχουν τώρα πολλοί που επενδύουν στον τομέα της γεωργίας και θα πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και να εξαιρέσουμε βέβαια αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη γεωργία για να εισπράττουν ε, πληρωμές και επιδοτήσεις. Κυρία Σένρα, ασχολήθηκα με τους νέους γεωργούς και αναφέρθηκα και με την διαγενειακή ανανέωση, αν θέλετε. Θέλουμε εμείς εκ των προτέρων να βοηθήσουμε οικονομικά τους νέους και στον τομέα της διαχείρισης και στον τομέα και τη στιγμή της κληρονομιάς και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με έναν τρόπο που θα στηρίξει τους νέους γεωργούς και για την ανάπτυξη της υπαίθρου τα μέτρα βοήθησαν και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία για την τροποποίηση των πολιτικών και των προγραμμάτων ιδιαίτερα μετά από ατυχή συμβάντα όπως οι μεγάλες πυρκαγιές οι οποίες ε, συνέβησαν. Βοηθήσαμε λοιπόν και στα πλαίσια της διαχείρισης ε, των δασών και της δασοκπονίας ε, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε τα ζώα να βόσκουν κάτω από τα δέντρα για να μην υπάρχει ευκολία στις πυρκαγιές των δασών. Γενικότερα υπάρχουν πολλά θέματα στη διαχείριση. Τώρα σε σχέση με τις τιμές, από τα μέσα του προηγούμενου χρόνου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 50% στις περισσότερες χώρες για τα γεωργικά προϊόντα και το ίδιο ισχύει και στην Ισπανία. Και έχετε δει τι έγινε με τις τροποποιήσεις στην συνδεδεμένη ε, βοήθεια ε, για τη Γαλλικία στο τομέα των γαλακτοκομικών. Ξέρω πως είστε κατά του εμπορίου και εκεί δεν θα συμφωνήσουμε. Όμως πρέπει να πω ότι εμείς ε, έχουμε αλληλεγγύη για την Αφρικανική Ένωση και από την πρωτοβουλία μου του Νοέμβριου του 2015 στη Βαλέτα, στην Σύνοδο Κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης, τοποθετήσαμε στο έγγραφο ένα κείμενο το οποίο καλείται, με το οποίο καλείται ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις ρίζες ε, του κακού που προκαλούν το φαινόμενο και οδηγούν τους ανθρώπους στη μετανάστευση ε, προς την Ευρώπη. Πολλές φορές οι μεσογειακές χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και ξέρετε πως κάθε χρόνο έχουμε 3,4 δις ε, ευρώ αγαθά να μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την, Ευρω... Ε, από την Αφρική, γεωργικά αγαθά, τα οποία δεν υπόκειται σε δασμούς. Εντάξει, εσείς μπορεί να μην θέλετε να έρθουν ε, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, αλλά το έχουμε συμφωνήσει και ε, στο Ναϊρόμπι το 2015 καταργήσαμε όλες τις εξαγωγικές πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθήσουμε την Αφρική. Και η Ευρώπη ε, ε, εκεί ηγήθηκε αυτής της προσπάθειας. Βλέπω πως δεν το γνωρίζετε. Αν είχατε διαβάσει τα έγγραφα θα τα ξέρατε αυτά. Κύριε Χόσλινγκ, ούτε εσείς διαβάσατε τα έγγραφα. Έτσι δεν είναι. Γιατί αν είχατε διαβάσει την ανακοίνωση θα διαβάζατε πως έχω εξηγήσει πως δεν πρόκειται να επανεθνικοποιήσουμε την γεωργία και θα μπορούσατε να το διορθώσετε αν το είχατε διαβάσει σωστά. Και δεν θα είμαστε λιγότερο φιλόδοξοι, θα είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι για το κλίμα και για το περιβάλλον. Νομίζω ότι πάρα πολλοί από τότε που έγινε εγώ επίτροπος και κάποια ακόμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εσείς οι ίδιοι που συνέχεια καταγγέλλεται το πόσο περίπλοκη είναι η πολιτική μας. Το λένε οι γεωργοί, το λένε τα κράτη-μέλη, το λέει το ελεγκτικό συνέδριο και καταγγέλει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε την περιβαλλοντολογική ε, πολιτική. Και δεν μπορώ να πιστέψω πως κάποιος θα μου πει πως η περιβαλλοντολογική πολιτική έτσι όπως εφαρμόζεται σήμερα θα πετύχει τους στόχους το 2030. Οπότε αυτό που γίνεται σήμερα δεν λειτουργεί. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να βρούμε άλλους τρόπους και να βασιστούμε στην εμπειρία της Γερμανίας και να δούμε πώς μπορούμε να προσφέρουμε μια ευκαιρία στο να επηρεάσετε και εσείς αυτέ τις πολιτικέ με έναν τρόπο που είναι πιο κατάλληλες για τι γερμανικέ συνθήκε. Θα έχει την ευκαιρία να το κάνει και η Ελλάδα και η Πορτογαλία και οποιοδήποτε άλλο κράτη-μέλη. Α ακούσουμε τι θέλουν τα κράτη-μέλη και για του περιβαλλοντικού στόχου και να δούμε τι θα γίνει, γιατί βέβαια αυτά θα τα επικυρώσει και θα τα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, επαναλαμβάνω, η πολιτική μα είναι κοινή γεωργική πολιτική και έχει στόχους για όλους και για τη βιοπικιλότητα. Αναφέρεται και αυτό συγκεκριμένα στην ανακοίνωση που έχω μπροστά μου. Και γίνεται και μια άμεση αναφορά στην σελίδα 24 σε πιο υγιεινό τρόπο διατροφής έτσι ώστε να μην έχουμε ε, τέτοια προβλήματα με την παχυσαρκία όπως επίσης ε, και με τα προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη ε, με την έλλειψη θρεπτικής διατροφής. Τώρα, για τα προβλήματα τα οποία αναφέρατε και εσείς κυρία μου, έχουμε μια ευκαιρία ε, να προσφέρουμε φαγητό υψηλής ποιότητας. Αλλά έχουμε και την ευκαιρία να εξάγουμε τα προϊόντα αυτά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέσεις απασχόλησης, δουλειές, απασχόληση στην Ήπεθρο. Διαφορετικά, ε, μόνο με τις τοπικές αγορές, αν δεν ε, εμπορεθούμε με τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν φτάνει. Κύριε Ραζούμ, Προσπαθούμε να εμπλέξουμε περισσότερο ε, τα κράτη-μέλη έτσι να μειώσουμε το φόβο των επιθεωρήσεων και των ελέγχων που έχουν αντιμετωπίσει οι Γεωργοί. Γιατί ναι, κάποιοι πραγματικά φοβόντουσαν και νομίζω πως ο κύριος Αντρέο και ο κύριος Οντέ και εσείς το έχετε θέσει σε πολλές περιπτώσεις και ο κύριος Ντεκάστρο. Οπότε ναι, κάποιες από τι δικέ σα ανησυχίε απηχώ εδώ με ένα νέο μοντέλο που θα μειώσει τον αριθμό των κανόνων, των ελέγχων, τη συμμόρφωση ε, με τεχνολογία έτσι ώστε να μην πηγαίνουμε στι εκμεταλλεύσει για να ελέγξουμε. Είναι πολύ επαγγελματικό αυτό το βήμα και επικοδομητικό και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις ρίζες του φαινομένου της μετανάστευσης, ας το αντιστρέψουμε και ας πούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία που έχουμε στη Γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ των Γεωργών στην Αφρική. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να συντονιστούμε καλύτερα. Το 60% των ανθρώπων στην Πεθρό, στην Αφρική, βασίζονται ε, για να επιβιώσουν στη Γεωργία. Να τους βοηθήσουμε λοιπόν να μείνουν στην Αφρική, να μην έρθουν στην Ευρώπη. Αυτό θέλει η πολιτική μας. Και βεβαίως νομίζω ότι σε πολιτικό επίπεδο θα συμφωνήσετε και περιμένω βέβαια να μην στηρίξετε και όλο στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Όπως σας είπα, θα συνεχίσουμε με μια άλλη σειρά ερωτήσεων. Ένα λεπτό. Ο κύριος Δεκάστρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Να του πω από την αρχή ότι εγώ διάβασα το έγγραφο. Και νομίζω δεν έχω την ανησυχία την οποία έχουν οι συνάδελφοι για τον κίνδυνο επανεθνικοποίησης. Είπατε Επίτροπε ότι η ΚΑΠ είναι μια επιτυχής διαδικασία. Και συμφωνώ μαζί σας. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι οι πάρα πολλοί γεωργοί είναι δυσαρεστημένοι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πάρα πολλοί γεωργοί στο Ηνωμένο Βασίλειο υπερψήφισαν το Brexit λόγω της περιπλοκότητας της ΚΑΠ. Και εάν η δήλωσή σας, εάν η δήλωσή σας σημαίνει ότι θα αλλάξουμε το παράδειγμα που προτείνουμε από μία Ευρώπη κυρώσεων σε μία Ευρώπη κινήτρων που προωθεί τις, την αριστεία, που προωθεί τις πρακτικές που ευνοούν το περιβάλλον και που δεν περιορίζεται στο να επιβάλλει κυρώσεις σε αυτούς που δεν υπακούν, τότε θα συνεργαστούμε σωστά. Είναι μια καλή βάση γιατί τότε θα έχουμε μια πραγματική νέα ευρωπαϊκή πολιτική που έχει σαν κέντρο τους γεωργούς. Εμεί νομίζω βοηθήσαμε ότι και με τον Ντατά και με τον ΤΕΣ βοηθήσαμε ιδιαίτερα για το Όμνιμπους τα θέματα στα οποία αναφέρεται, δηλαδή νέοι γεωργοί, αυξήσαμε τη βοήθεια, διαχείριση της, του κινδύνου μέσα από καταλληλότερα μέσα, ενίσχυση των γεωργών κτλ. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε ένα επιπλέον βήμα και εγώ έχω την άποψη ότι μπορούμε να εργαστούμε σωστά, αλλά να μην ξεχνάμε ότι με το Omnibus χρειαστήκαμε 15 μήνες από τη στιγμή που κατατέθηκε η πρώτη πρόταση και το πετύχαμε. Ελπίζω λοιπόν στα πλαίσια της ανακοίνωσης αυτής να λάβετε υπόψη τη συζήτηση η οποία υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, να υπάρξει μια νομοθετική πρόταση. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώσουμε όμως την διαδικασία. Ευχαριστώ. Επίτροπε, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η νέα αγροτική πολιτική θα είναι δίκαιη και ότι θα προσφέρει ισορροπημένες και δίκαιες συνθήκες για όλους τους αγρότες, όπου και αν βρίσκονται. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε και μία δίκαιη κατάσταση όσον αφορά τις τιμές. Κοιτάξτε πώς ήταν ε, στη Λιθουανία το φθινόπορο και κοιτάξτε πώς είναι σήμερα. Βλέπετε τι χρησιμοποιούν, ποιος είναι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στα λιβάδια και στα δικά μας ε, χωρίς ε, αλληλεγγύη, χωρίς την ευρωπαϊκή στήριξη δεν μπορούν να επιβιώσουν οι αγρότες μας. Πιστεύω ότι και στη Λιθουανία, η, στη γειτονική μας χώρα, θα στηρίξουν τους γεωργούς και ότι η νέα αγροτική πολιτική θα μπορέσει να δώσει τα εργαλεία για να διαχειριστούμε την κρίση. Η Πορτογαλία θα γνωρίσει μία από τις πιο σοβαρές κρίσεις λόγω της ξηρασίας. Είχαμε πυρκαγιές και φυσικά η ξηρασία είναι κάτι που έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την δουλειά των γεωργών μας. Δεν υπάρχουν βοσκοτόπια, και αν δεν βρέξει η συγκομιδή του 2018 θα είναι άθλια. Χρειάζονται έκτακτα μέτρα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την έκτακτη κατάσταση. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να θίξω. Το δεύτερο, όσον αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό της κοινή αγροτικής πολιτικής. Δεν πιστεύετε ότι κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση με σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου θα υπάρχει αγροτική πολιτική, η οποία δεν θα είναι όμως κοινή. Είναι τόσο περίπλοκη η υλοποίηση, τόσο περίπλοκη η έλεγχη. Δεν νομίζετε ότι αυξάνεται τη γραφειοκρατία για τους γεωργούς και δεν την απλοποιείτε. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της επικουρικότητας. Μπορείτε να μας δώσετε συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς προτίθεστε να μειώσετε το χάσμα μεταξύ των κρατών μελών, τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Επαναλαμβάνετε ότι θα ολοκληρώσετε και δεν ολοκληρώνετε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι μια καλή βάση για τη μελλοντική πολιτική μας. Προτείνεται λύσεις για την απλοποίηση της κοινή αγροτικής πολιτικής και να μειωθεί το γραφειοκρατικό άχθος για τους αγρότες. Χαιρετίζουμε την προσέγγιση σας όσον αφορά την ανακατανομή των ε, άμεσων πληρωμών, ένα μέτρο πολύ πιο ισορροπημένο για άμεσες ε, πληρωμές δεν θα φτάνουν μόνο στις ε, μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Βεβαίως καταλαβαίνουμε και τον στόχο για να τεθεί ένα όριο στις άμεσες πληρωμές και να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στους μικρούς γεωργούς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν διακρίσεις μεταξύ των νέων γεωργών και των γεωργών που ξεκινούν αυτή τη δραστηριότητα. Είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες γεωργών. Επίσης, το θέμα των δανείων και των πιστώσεων και του μηχανισμού που θα εναρμονίσει την παροχή δανείων στους νέους γεωργούς. Πώς διασφαλίζεται ότι η αγροτική πολιτική θα παραμείνει κοινή. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει περάσει τόσος χρόνος από τότε στην Επιτροπή μας συζητήσαμε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για την περίοδο 2005-2013. Είναι μια περίοδος βέβαια πριν αναλάβετε εσείς τις ευθύνες της γεωργίας, αλλά στην έκθεση αυτή είχαμε διαβάσει πως υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές αρνητικές τάσεις. Η πρώτη είναι η μείωση στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων. Χίλιες εκμεταλλεύσεις την ημέρα χάνονται και είναι κυρίως οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Και το άλλο είναι βέβαια ότι η γυράς και ο πληθυσμός των γεωργών, το 80% των γεωργών στην Ευρώπη είναι 45 και πάνω. Αν λοιπόν αυτές οι δύο διαδικασίες, μάλλον αυτές οι δύο τάσεις συνεχίσουν έτσι, η ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη θα κινδυνεύσει. Δεν θεωρείτε λοιπόν κι εσείς κύριε Επίτροπε πως η ΚΑΠ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αναστρέψει τέτοιου είδους τάσεις και επίσης δεν φτάνει η ΚΑΠ. Μήπως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε και κάποια κονδύλια από την πολιτική συνοχής. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ διάβασα την έκθεση, κύριε Πίτροπε, και στη σελίδα 14 πολλοί από εμάς πραγματικά μείναμε άφωνοι από τα στοιχεία που έχουν στο γράφημα με τη διαφορά μεταξύ γεωργικού εισοδήματο ε, στα κράτη-μέλη και βέβαια τη διαφορά που έχει το εισόδημα αυτό από το εισόδημα που αποκτάται από βιομηχανικέ δραστηριότητες. Στη χώρα μου η διαφορά αυτά είναι γύρω το 1 τρίτο, ε, είναι, είναι κατά 2 τρίτα χαμηλότερο. Δηλαδή οι γεωργοί ε, έχουν εισόδημα που είναι το 1 τρίτο αυτών που δουλεύουν σε άλλους τομείς. Άρα λοιπόν πώς θα τους παροτρύνουμε να συνεχίσουμε να εργάζονται στις εκμεταλλεύσεις τους. Δεν πρόκειται οι κοινότητες υπαίθρου να επιβιώσουν με τον τρόπο αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι καταρχήν είναι καλύτερε οι τιμές για τα προϊόντα τους και δεύτερον πώς θα κατευθύνουμε ε, την απαραιτητε τις απαραίτητες ε, στηρίξεις και επιδοτήσεις στα άτομα που χρειάζονται περισσότερο και στη διαρροή που Ε, στη διαρροή της ε, ανακοίνωσης ε, είχαμε, είχαν προταθεί από την Κομισιόν κάποια ανώτατα όρια. Δηλαδή δεν θα μπορεί κανείς να εισπράττει επιδοτήσεις πάνω από 100.000 ευρώ. Αυτό ήταν το όριο. Κάτι το οποίο δεν βρίσκουμε πια στην ανακοίνωση. Άρα λοιπόν κύριε Επίτροπε θα συνταχθείτε μαζί μας, θα προσπαθήσετε κι εσείς να γίνει πιο δίκαιη η ΚΑΠ έτσι ώστε να μην έχουμε αυτή τη γελία κατάσταση που ένα πολύ μικρό κομμάτι του γεωργικού πληθυσμού λαμβάνει το μερίδιο του λέοντα των επιδοτήσεων, ενώ οι άλλοι ε, κάθε μέρα αγωνίζονται για να τα καταφέρουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε και εγώ ε, καλωσορίζω την ανακοίνωσή σας. Είστε καλή. Και είναι και ενδιαφέρουσα, γιατί πιστεύω πως είναι καλύτερο να έχουμε μια πολιτική που βασίζεται στο να παραδίδει τα επιδιωκούμενα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι αυτό που έχουμε σήμερα είναι μια ε, προσέγγιση που μπορεί να μετρηθεί μεν, αλλά το κουστούμι που έχουμε κόψει δεν ε, μπορεί να το φορέσει κανείς. Ε, γιατί το αποφασίζουμε στις Βρυξέλλες χωρίς να ζητήσουμε τη γνώμη των κρατών μελών. Αλλά αν εσείς μπορείτε να μας βρείτε ένα σύστημα που είναι καλύτερο από την πολλαπλή συμμόρφωση, από το πρασίνισμα, από ε, τις ερεσιμότητες και έτσι να έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα είναι κατάλληλος για το στόχο του, fit for purpose, τότε ναι και θα έχουμε καλύτερα παραδοτέα και θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα δίνει κίνητρα και δεν θα επιβάλλει κυρώσεις. Αλλά η ερώτηση μου είναι έχουμε καταφέρει κάτι τέτοιο. Με ποιο τρόπο λαμβάνουμε εδώ υπόψη την εμπειρία και τα διδάγματα που έχει αποκομίσει ο ίδιος ο παραγωγός πώς αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη να πετύχουν τους στόχους τους, χωρίς να τους προγραμματίζουμε εμείς ε, ε, και σε εθνικό επίπεδο, όχι μόνο στο δικό μας επίπεδο. Θα πρέπει οι ίδιοι οι γεωργοί να αποφασίζουν ποια είναι τα μέτρα που χρειάζονται, γιατί αυτοί γνωρίζουν περισσότερο ποιες είναι οι ανάγκες τους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Χόγκαν. Η κοινή αγροτική πολιτική είχε πολλά θύματα τα τελευταία χρόνια και όλες οι οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες ε, καταραίουν ε, κάτω από το βάρος των ε, κανονισμών και των απαγορεύσεων. Μας είπατε κύριε Επίτροπε ότι Φυσικά και ασχολήθηκατε και με την ευημερία των ζώων. Όμως αν βγάλουμε τον τίτλο, μόνο σε δύο σημεία αναφέρεται η λέξη αυτή η ευημερία των ζώων. Πότε επιτέλους θα κάνει κάτι συγκεκριμένο η Επιτροπή, τι θα κάνετε. Δεν αναφέρεστε στην χρηματοδότηση για την τήρηση των κανόνων που αφορούν την ευημερία των ζώων. Λέτε ότι έχετε μια πιο βιώσιμη προσέγγιση, αλλά δεν βλέπω κάτι τέτοιο στις προτάσεις σας. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, μας μιλήσατε για απλοποίηση, για εξυγχρονισμό, μιλάτε για υποχρέωση αποτελεσμάτων και λέτε βεβαίως ότι είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Κοιτάξτε όμως ε, ποιος είναι ο ορισμός και τι ακριβώς αναθέτεται στα κράτη-μέλη. Η Ευρώπη θέτει στόχους περιβαλλοντολογικούς και η υλοποίηση αναπόκειται στα κράτη-μέλη. Αυτό σίγουρα θα οδηγήσει σε περισσότερο κατακαιρματισμό στην ενιαία αγορά. Κύριε Επίτροπε, περιμέναμε κάποια εργαλεία για τη διαχείριση των κρίσεων, αντιμετώπιση των κινδύνων. Είδατε τις εκθέσεις μας, τα συμπεράσματα της Task Force και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις στον προϋπολογισμό της κοινή αγροτικής πολιτικής. Οι γεωργοί δεν αντέχουν άλλες αλλαγές. Κάθε τρία χρόνια αυξάνοντας τη σύγχυση και μειώνοντας τις δυνατότητες να βρεθούν λύσεις. Ας κρατήσουμε λοιπόν την αγροτική πολιτική που είναι η μόνη πραγματικά κοινή πολιτική. Μια πολιτική που προσφέρει υγιή και ποιοτικά είδη διατροφής στους Ευρωπαίους πολίτες. Πραγματικά Έχω απογοητευτεί, διότι λείπει το όρομα από την παρουσίασή σας. Ο κύριος Γιάρα. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Ναι, μιλάτε για περισσότερη ευελιξία, αυτό είναι πάρα πολύ ελκυστικό, στόχοι, προσανατολισμένοι στόχοι, προϋποθέσεις. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε να μην υπάρξει περισσότερη σύγχυση στα κράτη-μέλη. Μιλάτε για τη μείωση της γραφειοκρατίας, για την απλοποίηση και λέτε ότι όσον αφορά το πακέτο των μέτρων, Υπάρχει το πρασίνισμα, το greening και υπάρχει μια ολόκληρη σειρά μέτρων που αναφέρονται στο δεύτερο πυλώνα. Βοηθήστε μας όμως να ενισχύσουμε τον πρώτο πυλώνα. Αυτό περιμένουν οι γεωργοί στην Ευρώπη. Εάν δεν υλοποιηθούν οι στόχοι, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ποιες θα είναι οι κυρώσεις για τα κράτη-μέλη. Εγώ σας προτείνω να υπάρξει μια πιο ίση κατανομή των άμεσων πληρωμών. Ναι, αναφέρεστε και εσείς αυτό. Το θέμα είναι εάν σε ένα κράτος μέλος ένας συγκεκριμένος αγρότης με 70 εκτάρια παίρνει άμεση πληρωμή ίση με αυτή που παίρνει ένας γεωργός με 600 εκτάρια σε ένα άλλο κράτος μέλος. Πού είναι η ίση κατανομή. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και νομίζω ότι θα πρέπει και εσείς να ακούσετε τις προτάσεις μας, να ακούσετε τις τροπολογίες μας και να ενσωματωθούν αυτά και να συμπληρώσουν τη δική σας πρόταση. Πρόεδρος, θα δώσω το λόγο στην κυρία Σράιερ. Ευχαριστώ. Είμαι ευτυχής για την πρότασή σας Επίτροπε. Γνωρίζετε όμως ότι ποτέ δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε πλήρως. Οι γεωργοί θα παραμείνουν γεωργοί, θα πρέπει να υπάρξουν όμως κάποιες ρυθμίσεις στον τομέα του περιβάλλοντος, οι οποίες ακόμα εκκρεμούν. Η διοπικιλότητα είναι με μια εθνική αρμοδιότητα, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ακριβώς το τι προτείνεται σε σχέση με αυτό. Τώρα για τους δικαιούχους το 80% ε, το παίρνει το 20%. Ε, είπατε ότι υπάρχουν ανώτατα όρια, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν χιλιάδες γεωργοί οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν ανώνυμες εταιρείες και να διατηρήσουν με τον ένα τρόπο ή τον άλλο τις επιδοτήσεις. Κύριε Επίτροπε, το θέμα της επικουρικότητας. Διαρωτώμε λοιπόν σε σχέση με την ε, ευελιξία. Αυτό σημαίνει... Και συγχρηματοδότηση, μήπως είναι μια ανοιχτή πόρτα εδώ στην επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ. Μια άλλη ερώτηση τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη ε, και να είναι πλέον διαφανή. Αν δεν πετύχουν τους στόχους αυτούς όμως, το τέλος ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, το κράτος μέλος ή η Γεωργία. Ποιος θα επιβάλλει την κύρωση, το κράτος μέλος ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ή θα τιμωρηθεί το κράτος μέλος. Και αυτό τι σημαίνει, απώλεια ε, εσόδων για το κράτος, για τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους. Και θα θέλατε να μου πείτε επίσης τι γίνεται με τις αναδιανεμητικές πλήρωμες. Ε, θα ήθελα να μάθω ακριβώς πού υπάρχει αναδιανομή, αναδιανεμητική λειτουργία, ανάμεσα σε ποιους, ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ε, στο εσωτερικό του, κάθος, του κάθε κράτους μέλους. Η ιδέα είναι πάρα πολύ δύσκολη για μένα σε σχέση με την μετανάστευση. Υπάρχει ένα θέμα δημογραφικό, αλλά εμείς πιστεύετε ότι μέσω της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου θα πρέπει να καλύψουμε ανάγκες για πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από εντελώ διαφορετικές πηγές, όπως η συνεργασία για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, λέει ο κύριος Καλινόφσκι. Νομίζω ότι σε πάρα πολλά σε πάρα πολλές συναντήσεις και από πάρα πολλούς εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλων των επιπέδων ακούμε συνέχεια πως υπάρχει θέμα ερεσιμότητας, πως θα πρέπει η αιρεσιμότητα να υπερισχύει τη στιγμή της πρόσβασης στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι γεωργοί θα πρέπει να πληρώσουν ε, τα σπασμένα γιατί κάποια κυβέρνηση ε, παραβιάζει τα, τους κανόνες μας. Νομίζω ότι είναι ανησυχητικό κάτι τέτοιο και φαντάζομαι ότι και εσείς θα είστε κατά ε, μιας τέτοιας προσέγγισης. Και έχω και μια δεύτερη ερώτηση τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή έχουν ένα βαθμό ευελιξίας. Για παράδειγμα, μπορούν να μεταφέρουν κονδύλια ανάμεσα στους δύο πυλώνες. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι περιορισμοί. Έχει να κάνει με την ίδια άζουσα κατάσταση κάποιες περιφέρειες κάποιας χώρας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια καλή λύση και θα ήθελα να μου πείτε ε, τι ακριβώς θα συμβεί με αυτή τη δυνατότητα και περιμένουμε βέβαια και τις νομοθετικές σας ε, προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία... Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ενδιαφέρουσα η πρότασή σας, ενδιαφέρουσα. Και είναι μια ευρεία ματιά. Αλλά έχω κάποια θέματα που εμένα μου δημιουργούν ερωτηματικά. Περισσότερη επικουρικότητα. Ναι, στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ανησυχώ για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, ποιες είναι οι επιπτώσει στην εσωτερική αγορά αυτής τη επικουρικότητα, γιατί υπάρχουν κοινοί κανόνες αλλά και μεγάλες διαφορές. Και δεύτερον, συγχρηματοδότηση ανοίγει αυτή η δυνατότητα. Και ανησυχώ, γιατί η επικουρικότητα αυτή δεν περιγράφεται παρκώς. Θα ήθελα να έχετε κάνει και κάποιες αλλαγέ τα εργαλεία ε, που χρησιμοποιείτε για να διαχειρίσετε τις, αγοράς, τις αγορές, τις ΚΟΑ και τα λοιπά, γιατί υπάρχουν βέβαια οι κανόνες για τους αθέμητους ανταγωνισμούς και τα λοιπά και στο ε, πολυνομοσχέδιο έχουν ενταχθεί κάτι τέτοιες ε, διατάξεις, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πώς θα εφαρμοστεί αυτό και τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ εγώ θα ζητήσω από την Ισπανία να κάνει μια παραπάνω προσπάθεια. Αλλά θα πρέπει εσείς να πείστε και τον Επίτροπο κύριο Έτιγκερ πως χρειάζεται περισσότερους πόρους. Αλλά οι περισσότεροι πόροι δεν θα πρέπει να ε, προέλθουν από την ΚΑΠ και από τα Ταμεία Συνοχής. Να προσπαθήσουμε εμείς ο καθένας να πει σε αυτόν που μπορεί. Και μια τελευταία ερώτηση. Τον Ιούνιο μπορούμε να εγκρίνουμε αυτές τις νομοθετικές προτάσεις χωρίς να υπάρχει το χρηματοδοτικό πλαίσιο, χωρίς να έχει εγκριθεί, γιατί θα εγκριθεί το Μάρτιο του 19. Πιστεύετε πως είναι εφικτό. Εγώ νομίζω ότι εσείς ναι. Έχετε, έχετε μεν όρεξη, αλλά τελικά τι έγινε με τη βιολογική γεωργία. Μας έμεινε η κληρονομιά από την προηγούμενη θητεία και πήρε τρία χρόνια να εγκριθεί. Ξέρω πως εσείς θέλετε να περάσει τον Ιούνιο, αλλά νομίζω πως είναι αδύνατον. Ευχαριστώ. Euh. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την παρουσίαση που μας κάνατε. Υπάρχουν κοινά σημεία με την οδηγία πλαίσιο για το νερό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες ανησυχίες που νομίζω ότι δικαιολογούνται όσον αφορά τη χρηματοδότηση και όσον αφορά την υλοποίηση. Στην τελευταία ΚΑΠ είχαμε προετοιμάσει καταπληκτικές προτάσεις. Όταν όμως έφτασαν για υλοποίηση, όταν δηλαδή τα κείμενα επεξεργάστηκαν από τις υπηρεσίες και άρχισαν να μπαίνουν στις λεπτομέρειες της χρηματοδότησης και της ανάκτησης κάποιων ποσών, η υλοποίηση ήταν πολύ διαφορετική. Άλλες διευθύνσεις από τη δική σας λοιπόν τελικά έχουν άποψη και επεμβαίνουν στις προτάσεις των κρατών μελών. Η πολιτική που αφορά το περιβάλλον, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τις απαραίτητες εγγύσεις έτσι ώστε να παραμείνει αυτό το έγγραφο, έγγραφο κυρίως που αφορά τη γεωργία. Αν θέλουμε να σκεφτούμε για το πλαίσιο, θα πρέπει να δούμε τι κάνουν και άλλοι. Υπάρχουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Εκπλήσωμαι γιατί στο κείμενό σας δεν αναφέρετε τίποτα για τα εργαλεία που θα καλύψουν την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου τη διαχείριση των κρίσεων. Μας είπατε ότι η διαχείριση της κρίσης θα γίνει στην επόμενη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής. Εδώ όμως δεν βλέπω τίποτα από αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Βέβαια, πρέπει να διαβάσουμε όλη την έκθεση για να δούμε όλες τις λεπτομέρειες των προτάσεών σας. Όσον αφορά τώρα τις πληρωμές για τις, τις άμεσες πληρωμές και την συνιστόσα του greening, του πρασινίσματος. Μπορείτε να μας πείτε ακριβώς τι θα παραμείνει στα κράτη-μέλη. Εγώ ξέρω ότι για την Ελλανδία τουλάχιστον τα προγράμματα συνεχίζουν να έχουν μια τέτοια συνιστόσα και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το κομμάτι του περιβάλλοντος. Δεύτερον, το θέμα της ευθύνη των αρμοδιοτήτων. Διαρκώς διαμαρτυρόμαστε προς την Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη λένε ότι έχει υπερβολικά σημαντικό έλεγχο η Επιτροπή επί της πολιτικής τους. Εδώ βλέπω ότι δίνεται κάποιες αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν θα αναλάβουν τις ευθύνες του τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, πώς καθορίζουμε το τι είναι ένας πραγματικά ενεργός γεωργός. Αυτό είναι ορισμός ε, της ΦΑΟ. Εγώ διάβασα πολύ προσεκτικά το έγγραφο και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ακριβώς ε, πώς ορίζονται οι εκμεταλλεύσεις ή τα άτομα που εργάζονται εκεί και πώς θα υπολογίζονται οι άμεσες πληρωμές. Είναι καλό να βλέπει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ασχολείται με θέματα όπως η φορά και άλλα θέματα τα οποία είναι σημαντικά για την οικονομία όπως η, ε, κυκλική η κύκλικη οικονομία, η, ε, η απασχόληση των νέων. Είναι λοιπόν θέματα σημαντικά για το μέλλον. Τώρα, διαχείριση των κινδύνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας δώσει εγγυήσεις έτσι ώστε οι ίδιες στρεβλώσεις της αγοράς να μην καταστήσουν μη βιώσιμη την, πολιτική, την παραγωγή της στην Γεωργία. Τώρα, σχετικά τώρα με την χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση των άμεσων πληρωμών. Αυτό δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στην τελική πρόταση. είναι το, ποια είναι η λύση γι' αυτό εμείς στην ανάπτυξη της υπαίθρου θέλουμε μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πολιτικές έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε την χρήση ε, των πιστώσεων. Ε, προτείνουμε μηχανισμούς έτσι ώστε να συνδυάσουμε και τις παρεμβάσεις από άλλες πολιτικές της κοινότητες της Υπέθρο. Ο μηχανισμό αυτός πώς προβλέπεται να λειτουργήσει. Ευχαριστώ, χαίρομαι που έχουμε τόσο κόσμο εδώ. Ε, συνήθως είναι άδεια η αίθουσα, τώρα φαίνεται ότι κάτι σημαντικό συμβαίνει. Ε, λέτε ότι τα μέσα και οι δράσεις για τα ανώτατα όρια και τη σύγκληση υπάρχουν ήδη και αναφερθήκατε ε, στις προτάσεις της υπόλοιπες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, προστασία του εισοδήματος και την προστασία επίσης και στήριξη της περιβαλλοντικής φιλικής, μάλλον για το περιβάλλον γεωργίας. Οπότε τι εμποδίζει να εφαρμόσουν τους κανόνες αυτούς οι εθνικές κυβερνήσεις όπως το έχει κάνει ή δεν το έχει κάνει η κυβέρνηση στην Ιρλανδία. Ε, κάθε χρόνο, σύμφωνα με το παλιό σύστημα, χρειάζονται συνεχώς επιπλέον χρήματα για να στηριχθούν, υποτίθεται, ε, τα αγροκτήματα και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στα θέματα της απασχόλησης. Δυστυχώς τίποτα δεν έχει γίνει. Κάποιες φάρμες θα πάρουν 700 ευρώ ανά εκτάριο και άλλες 168 Συνεπώς λοιπόν ε, τέτοιου είδους ε, συστήματα είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποτραπεί. Και τώρα οι πληρωμές για το greening θα παραμείνουν στον πρώτο πυλώνα και σχετικά με την ακρίβεια των εγγράφων σας. Λέτε εδώ και έχετε πει και ε, σε άλλες ευκαιρίες ότι οι πληρωμές βασίζονται στην επιφάνεια, στη γη. Δεν βασίζονται στην επιφάνεια εκτός ε, από τις ε, ε, χώρες οι οποίες έχουν flat rate πληρωμές. Συνεπώς λοιπόν δεν πρέπει να αναφέρεστε σε θέματα τα οποία δεν ισχύουν εδώ, στην χώρα μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, θα παραμείνουν οι πληρωμές για τον Greening στον πρώτο πυλώνα και τι θα εμποδίσει τις κυβερνήσεις να παραβιάσουν τους κανόνες αυτούς. Αγαπητέ, θα διαφωνήσω μαζί σας. Δεν είναι συνήθως άδεια η αίθουσα αυτή, μια φορά συνέβη. Σας παρακαλώ πολύ, μη γενικεύετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κάποια από αυτά που αναφέρετε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προτάσεις και νομίζω ότι υπάρχουν νέοι τρόποι, νέες απαντήσεις το θέμα των περιβαλλοντικών μέτρων που θα πρέπει να τα ξαναδούμε και να ξανασκεφτούμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Άλφρεντ αναφέρθηκε στις ε, προτάσεις σας και στις ανησυχίες που παρόλα αυτά συνεχίζουμε να έχουμε το ρόλο των κρατών, το ρόλο των διαφόρων μεγάλων και μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, ιδιαίτερα στον τομέα των οποροκυπευτικών. Όσον αφορά τώρα τον υπολογισμό των ε, άμεσων πληρωμών στη, στον πρώτο πυλώνα. Σήμερα ξέρουμε ότι καταβάλλονται ποσά και υπολογίζονται αυτά βάσει μιας ιστορικής, θα, θα λέγαμε, αξιολόγησης και βασίζονται σε κάποια δεδομένα πριν πολλές φορές από 27 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σε καμία περίπτωση, αν δεν μεταρρυθμιστεί, αν δεν αλλάξει, δεν μπορούμε ποτέ να μιλάμε για σύγκληση και δεν θα την πετύχουμε ποτέ αυτή τη σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είστε ένας ε, μικρομπακάλης. Α, βλέπω ότι μας κρύψατε κάποια πράγματα. Μας κρύψατε ένα έγγραφο που ήρθε εδώ πριν από μια εβδομάδα. Ήταν ένα έγγραφο το οποίο πραγματικά, από το οποίο έλειπαν κάποια σημεία, όπως το 4-2. Κύριε Πρόεδρε, δεν μας το ανέφερε. Είναι το πιο πολιτικό σημείο. Έλειπε από το έγγραφο. Και εδώ βλέπουμε ότι μιλάτε για μια βελτίωση της ε, κοινή αγροτικής ε, ε, πολιτικής με την ενσωμάτωση των μεταναστών. Μα αυτή είναι η βελτίωση. Μα αυτό είναι σκάνδαλο. Θέλετε να αντικαταστήσετε τους γεωργούς που αυτοκτονούν από τους μετανάστες. Μα αυτό είναι καθαρή αυτοκτονία πολιτική. Κύριε Επίτροπε, πραγματικά νομίζω ότι πάτε αντίθετα με αυτό που προσδοκεί ο λαός στην Ευρώπη. Όχι, δεν θέλουμε μετανάστες και δεν θέλουμε μετανάστες στην Ήπεθρο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πολλά έχουν να γίνουν ακόμα. Θα δώσω το λόγο τώρα στον επόμενο συνάδελφο. Η ανακοίνωσή σας δίνει κάποιε κατευθυντήριες γραμμές που θα δώσουν στους Ευρωπαίους Γεωργούς ε, ένα περιθώριο ανακούφιση. Όμως υπάρχουν πολλές διαφορές από την προηγούμενη εκδοχή. Η προηγούμενη εκδοχή έγραφε η ΚΑΠ θα πρέπει να συνεχίσει να μειώνει τις διαφορές μεταξύ των ε, επίπεδων στήριξη ανάμεσα σε κράτη-μέλη. Και αυτή τη στιγμή το κείμενο διαβάζει. Η ΚΑΠ θα πρέπει να μειώσει τι διαφορέ μεταξύ κρατών-μελών στο σε σχέση με το θέμα της στήριξης. Δεν νομίζω ότι εδώ είναι απλή ε, γραμματική αλλαγή, αλλά φοβάμαι ότι μέσω αυτής τη αλλαγή θα έχουμε πολλές συνέπειες. Θα πρέπει όλοι οι γεωργοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνουν την ίδιο επίπεδο χρηματοδότηση στα πλαίσια τη επόμενη ΚΑΠ σε αγοράζουμε και ακολουθούμε τους ίδιους νομοθετικούς κανόνες. Άρα θα ήταν άδικο να μην στηρίζονται τα κράτη-μέλη τα οποία ε, προσχώρησαν ε, το 4, το 7, το 13. Μπορείτε να δεσμευτείτε λοιπόν πως θα έχουμε ίση χρηματοδότηση για όλους, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για μια νέα νέου είδους ε, κοινή αγροτική πολιτική, θέτεται στόχους και μετά τα αναθέτεται στα κράτη-μέλη να τα υλοποιήσουν. Βεβαίως, ο καθορισμός των στόχων είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να δημιουργήσει πολλή ένταση. Μιλήσατε όμως για κάτι που δεν είναι και πολύ καινούριο, διότι στο δεύτερο πυλώνα έτσι και αλλιώ τα κράτη-μέλη έχουν πολλές αρμοδιότητες. Όσον αφορά τώρα το greening, το πρασίνισμα, εδώ βλέπουμε ότι δεν υλοποιούνται οι στόχοι, ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση. Έχουμε προβλήματα, έχουμε δυσκολίες και στον τομέα της βιοπικιλότητας και στον τομέα του περιβάλλοντος. Και δεν μπορούμε καν να μιλήσουμε σήμερα για κοινά πρότυπα, για κοινά θεμέλια πάνω στα οποία θα στηρίξουμε αυτή την πολιτική. Καθορίζεται λοιπόν στόχος, θέτετε δείκτες, κάνετε καλή καθοδήγηση, κάνετε καλή, δίνετε καλή κατεύθυνση, αλλιώς Εάν ανατεθούν όλα στα κράτη-μέλη, χωρίς επιτήρηση, χωρίς έλεγχος, ε, δεν υπάρχει καμία μεταρρύθμιση, καμία κοινή αγροτικής πολιτικής. Um, Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Μπράνεν. Καταρχήν, Λυπάμαι που έφτασα καθυστερημένα και έχασα την ομιλία σας, ε, κύριε Επίτροπε, αλλά ήμουνα, σε δύο, ήμουνα δύο ρόφους πιο ψηλά όπου συζητούσαμε τα θέματα της ε, δασοκομείας και εκεί πρέπει να σας πω πως το 19% των γεωργικών γεών καλύπτονται από δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν αναμειγνύουμε ε, ε, στη γεωργική γη δέντρα τότε τα αποτελέσματα είναι πραγματικά πάρα πολύ θετικά. Δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα, δεν έχεις πρόβλημα με τις πλημμύρες Θέλω να σας δείξω και ένα φυλάδιο ε, που μας δίνει 50 ε, παραδείγματα για το πώς η αγρό ε, δασοκομεία βελτιώνει το γεωργικό περιβάλλον στην Ευρώπη. Εσείς είπατε πως δεν θα επιβάλλει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση πόσα δέντρα μπορεί να έχει μία εκμετάλλευση στα χωράφια της. Νομίζω ότι θα σας κεράσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Μπορούμε λοιπόν εμείς οι δυο μας να κρίνουμε ότι μια κίνηση είναι πιο νόστιμη, καλύτερη γεύση αν το κρυθάρι το οποίο έχει οργωθεί σε ένα χωράφι που είχε και δέντρα είναι καλύτερης ποιότητας από ένα κρυθάρι, από ένα απλό χωράφι. Ε, νομίζω, λέει ο Επίτροπος, ότι άμα πίνουμε μια γκίνες μπορούμε να συζητήσουμε και θέματα πιο ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερο το έγγραφο το οποίο μας παρουσιάσατε. Σας ευχαριστώ για τη συνεχιζόμενη στήριξη προς τους γεωργούς. Ακούσαμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που είπατε και για τις άμεσες πληρωμές. Είπατε ότι είναι ένα δίκτυο ασφαλείας για τους γεωργούς. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες ε, λεπτομέρειες για τη γραμμικότητα των άμεσων πληρωμών. Εγώ ε, Διάβασα και αυτό το οποίο είπατε σε σχέση με την παρουσίαση ε, του κυρίου Γιούνκερ για την ισότητα Ανατολής Δύσης και Βορρά Νότου. Εδώ θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω ότι η κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να μειώνει τις διαφορές. Θα έπρεπε ή οφείλει να το κάνει. Γιατί πραγματικά εγώ ανησυχώ από τον γραμμικό χαρακτήρα των άμεσων πληρωμών ανάμεσα ε, στη δυτική και την ανατολική πλευρά της Ένωσης. Δεν πάβει η αγορά να είναι ταυτόσιμη, ανεξάρτητα από το πώς βλέπουμε λοιπόν ε, τις άμεσες πληρωμές, με ανώτατο όριο ή όχι, ε, θα πρέπει για όλες τις χώρες να ισχύουν τα ίδια, γιατί όλες οι χώρες πρωταγωνιστούν στην ίδια την αγορά. Μία ερώτηση θα ήθελα να θέσω και εγώ αν μου επιτρέπετε. Καταρχάς, στους κοινού στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη ε, προετοιμάζουν τον επαναπροσανατολισμό της στρατηγικής, έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους. Αυτή η στρατηγική θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από την Ευρωπαϊκή, Πολιτική, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς λοιπόν στο πλαίσιο αυτό θα διατηρήσετε τα κριτήρια τα οποία απαιτούνται, θα υπάρξουν συγκεκριμένες οδηγίες ε, για τους στρατηγικούς τομείς, ε, για την αμοιβαία αναγνώριση είναι κάτι το οποίο θα συνδεθεί με συμπληρωματικές εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας δώσετε κάπως περισσότερες ε, λεπτομέρειες, λέει ο Πρόεδρος. Επίτροπε, έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε μιλήσει αρκετά για την αγορά, έχουμε, δεν έχουμε μιλήσει για τη σταθεροποίηση, για τις κρίσεις και για τα εισοδήματα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τέλος, σχετικά με τις εξωτερικές αιρεσιμότητες, γιατί όλα τελικά επηρεάζουν την ΚΑΠ. Η ΚΑΠ αυτή ε, θα τεθεί σε λειτουργία από το 2021. Έχουμε λοιπόν αρκετά χρόνια μπροστά μας. Εν τω μεταξύ έχουμε μπροστά μας μόνο το Omnibus μέσο, το οποίο σίγουρα μπορεί φυσικά να, να απλουστεύσει, να διευκολύνει ορισμένα πράγματα για τους γεωργούς, και να καταστήσει την κοινή αγροτική πολιτική πιο εύπεπτη. Όλοι το έχουμε πει λοιπόν. Επιθυμούμε μία ισχυρή ΚΑΠ. Ξέρω ότι η κοινή αγροτική πολιτική δεν είναι μόνο πληρωμές, δεν είναι μόνο χρήματα, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Πώς θέλουμε εμείς να καλύψουμε ε, τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν σε οικονομικό επίπεδο από το Brexit. Πρέπει να πούμε στους γεωργούς ότι θα υπάρξουν λιγότερες πιστώσεις. Δεν αναφέρομαι σε νέες προκλήσεις. Μπορούμε να φανταστούμε ότι θα μπορούσε τις νέες προκλήσεις να τις χρηματοδοτήσει η πολιτική συνοχής. Όμως, όμως λέγω, αυτή η κοινή πολιτική είναι κοινή όχι μόνο λόγω των ευρωπαϊκών πιστώσεων, αλλά κυρίως λόγω της αγοράς της ενιαίας. Οπότε υπάρχουν πολλά τα οποία μένει να γίνουν. Και το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να καλύψουμε τα προβλήματα και τις ελλείψεις που θα, θα προκαλέσει το Brexit με εθνικές παρεμβάσεις, αλλά όχι με κοινοτικές παρεμβάσεις με παρεμβάσεις στον τομέα τον εθνικό. Μόνο και μόνο για να καλύψουμε τα ελλείμματα που θα δημιουργηθούν από το Brexit και να διατηρήσουμε μια κάποια ισορροπία. Είναι σαφές ότι οι πιο πλούσιες χώρες δεν πρόκειται να δώσουν περισσότερα χρήματα. Ξέρω ότι η συζήτηση αυτή δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς Κανένας δεν πιστεύει ότι τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο θα αυξήσουν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέσα για τη γεωργία. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά μερικές φορές θα πρέπει να συζητάμε ακόμα και τα δύσκολα, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ όλους όσους ε, έκαναν ερωτήσεις. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι σαν επίτροπος με αυτό το έγγραφο που συμπεριλαμβάνει και τα θέματα που αφορούν τον προπλήγμα. Θα πρέπει όμως οτιδήποτε αφορά αυτό το θέμα να περιμένετε μέχρι το Μάιο και θα σας δώσω πολύ περισσότερες πληροφορίες. Όπως ξέρετε δεν έχει αποφασιστεί ακόμα το θέμα του προπλήγματος και το θέμα των επιπτώσεων του Brexit επί του προϋπολογισμού. Έχουμε 10 με 12 δις λιγότερα. Είναι η άμεση συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου συνολικά στον προϋπολογισμό. Η μία εναλλακτική είναι να αυξηθεί η συνεισφορά των κρατών μελών για να καλυφθεί αυτό το κενό στον προϋπολογισμό. Δεύτερον, μπορεί να υπάρξουν και κάποιες νέες πρωτοβουλίες, μέσω των οποίων θα υπάρξει νέο φρέσκο χρήμα και βεβαίως εάν υλοποιηθεί εδώ η υλοποιηθούν διάφορες προτάσεις έκθεσης μάτι, εδώ μπορεί να υπάρξει αυτό το νέο χρήμα. Ή τρίτη αναλλακτική να υπάρξει περιορισμός των δαπανών. Αυτές είναι οι τρεις εναλλακτικέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι μπορώ να το επαναλάβουμε αλλά φυσικά και πέρα από την κοινή αγροτική πολιτική υπάρχουν και άλλοι τομείς ε, στους οποίους ισχύει αυτό που σας λέω. Τους τελευταίους έξι μήνες ακριβώς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να κοιτάξουμε όλες αυτές τις. Ο κύριος Δεκάσο και άλλοι μίλησαν για το πάρα πολύ σημαντικό θέμα της διαχείρισης του κινδύνου. Ναι, βάσει του κανονισμού Omnibus πολλά πολύ θετικά έχουν γίνει για το πώς μπορούμε να φτάσουμε σε ε, εργαλεία, μηχανισμούς σταθεροποίησης. Θα πρέπει να δούμε επίσης και για τις αρμοδιότητες των ενώσεων παραγωγών. Ε, λήφθησαν πολύ σημαντικές αποφάσεις, ε, παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, που αφορά το δίκαιο του ανταγωνισμού στο θέμα αυτό. Ναι, χρειάζεται να δοθεί περισσότερη έμφαση και στις εγγύσεις, αλλά και στην ασφάλεια, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν κάποιες επιπτώσεις της κρίσης και πραγματικά πιστεύω ότι εδώ πέρα από το οργανισμό Omnibus θα πρέπει να συνεχίσουμε. Υπάρχουν ε, βεβαίως κρίσεις εκτός της ΚΑΠ, κρίσεις εντός της ΚΑΠ, κρίσεις που επηρεάζουν την ΚΑΠ, όμως δεν είναι στο εσωτερικό της. Θα πρέπει να δούμε πώς όλα αυτά μπορεί να καλυφθούν. Μιλήσατε για την ξηρασία στην ε, Πορτογαλία, στην Ισπανία, πλημμύρες στη Φιλανδία, στις χώρες της Βαλτικής. Ναι, χρειάζεται ένδειξη αλληλεγγύης με όλες αυτές τις χώρες και με όλους αυτούς που πλήττονται. Και με μεγάλη επιτυχία βεβαίως το έχουμε κάνει. Παραδείγματο χάρη για τους σεισμόπληκτους την τελευταία φορά. Διαχείριση κρίσεων λοιπόν, ναι, διαχείριση κινδύνου. Εγώ είχα επισκεφθεί πρόσφατα την Πορτογαλία και ναι, βεβαίως και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την ξηρασία και θα τροποποιήσουμε τον κανονισμό για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Δεν έβρεξε για έξι μήνες. Εγώ όμως όταν πήγα έβρεχε. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα για να διασφαλίσουμε ότι όντως υπάρχει κάλυψη των αναγκών και προστασία. Ναι, θα απλοποιήσουμε την κοινή αγροτική πολιτική και θα υπάρξει κοινή αγροτική πολιτική με την μεταρρύθμιση. Φυσικά, το θέμα της σύγκλησης. Το θέμα της σύγκλησης είναι πολύ σημαντικό και αυτό βέβαια, όποια και να είναι η απόφαση, θα έχει θετικές επιπτώσεις και στην Πορτογαλία. Χρειάζεται καταρχήν η πρώτη απόφαση γενικά για τον προϋπολογισμό και βεβαίως να αυξήσουμε τα μέτρα που θα οδηγήσουν στη σύγκληση με μεγάλη χαρά. Αλλά εδώ σίγουρα θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Άλλα κρατημέλη θέλουν και άλλα δεν θέλουν. Αναφερθήκατε και στους νέους γεωργούς. Επί χρόνια νομίζω ότι τα μέτρα στήριξης των νέων γεωργών ήταν σημαντικά. Θα κάνουμε πολύ περισσότερα για αυτούς που θέλουν να εγκατασταθούν και βεβαίως να δώσουμε περισσότερα κίνητρα σε αυτούς που θέλουν να αποχωρήσουν έτσι ώστε να αναλάβει κάποιος τις επιχειρήσεις τους. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας και εδώ αλλά και έξω από αυτήν την αίθουσα. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε την απλή δημιουργία στόχων, θέση στόχων, αλλά να παρακολουθήσουμε και το τι γίνεται από εκεί και πέρα. Βεβαίως και για τους γεωργούς χρειάζεται στήριξη των ε, επενδύσεων, στήριξη της χρηματοδότησης και βεβαίως η έγκριση των προτάσεων αυτών από την Επιτροπή θα ελέγξει ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς στόχους και τους στόχους της μεταρρύθμισης της κοινή αγροτικής πολιτικής. Με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύσουμε το κοινό κομμάτι της κοινή αγροτικής πολιτικής. Σκοπός μας είναι βεβαίως να συνεισφέρουν περισσότερο οι αγρότες, περισσότερο τα κράτη-μέλη, αλλά να υπάρξει ευελιξία μέσω της επικουρικότητας να δράσουν και τα κράτη-μέλη. Και βεβαίω θα πρέπει τα κράτη-μέλη να επιλέξουν μέσω των στόχων που προτείνει η κοινή αγροτική πολιτική. Στην ε, Γερμανία, παραδείγματο χάρη, με τις, ε, τα κρατήδια και ο υπουργός ο κύριο Σμιτ, ο ομοσπονδιακό υπουργό, έχει να κάνει και με τους ε, αρμόδιους Υπουργούς Γεωργίας του κάθε κρατηδίου. Και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο υπάρχει συντονισμός με την κοινή αγροτική πολιτική. Αυτή είναι όμως, αν θέλετε, η φύση της πολιτικής μας. Βασιζόμαστε στην επικουρικότητα και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα πορευθούμε θέτοντας αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη και με τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους, όπως παραδέχαμε τους χάρη αυτό που στη Γερμανία. Τώρα, όσον αφορά το παρόν σύστημα του πρασινίσματος, του greening, θα αντικατασταθεί από ένα καινούριο. Ήταν πολύ περίπλοκο το σύστημα μέχρι τώρα, με διαφορετικά συστήματα αρισιμότητας, με καλές ε, βέλτιστες πρακτικές, με συμμόρφωση και πολλές πολλές επικαλύψεις. Χρειάζονται συστήματα ανάπτυξης της υπαίθρου και θα προσπαθήσουμε να απλοποιήσουμε τα συστήματα αυτά. Σήμερα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θέτουν τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στον τύπο της γεωργίας και των γεωργικών εκμεταλλευτών τους. Οπότε θα έχουμε ένα σετ ε, κανόνων για τη διαχείριση που θα πρέπει να ακολουθούν τα κράτη-μέλη και οι γεωργοί. Θα χρησιμοποιήσουμε δορυφορικά στοιχεία που θα μειώσουν το βάρος, δηλαδή σε ανθρώπινο δυναμικό για να ελέγχουν τους γεωργούς και βεβαίως και θα βελτιώσουν το κλίμα γύρω από τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους. Άρα λοιπόν θα μπορέσουμε να κάνουμε πάρα πολλά μέσω της τεχνολογίας. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξηγήσουν ποια είναι η βασική γραμμή πάνω από την οποία μπορούν να οικοδομήσουν και εθελοντικά μέτρα. Να μην έχουμε επικαλύψει, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται δύο έλεγχοι. Ένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ένα σε επίπεδο κρατών μελών. Οπότε θέλουμε να μειώσουμε, να εξορθολογήσουμε και από το 5% των ελέγχων να φτάσουμε στο 1% με δορυφορική τεχνολογία για το μεγαλύτερο ποσοστό αυτό αλλά θέλουμε και μεγαλύτερη φιλοδοξία για το περιβάλλον και το κλίμα. Σε τοπικό επίπεδο, καλύτερη στόχη για να πετύχουμε τις δεσμεύσεις μας και αυτό θα ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να κάνουν. Και βεβαίως θα τα εγκρίνει όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μου είπατε πολύ συχνά πως τα μέτρα που αποφασίζουν οι Βρυξέλλες δεν παραδίδουν αυτά που επιθυμούμε για το περιβάλλον. Θέλουμε περισσότερο. Και χρειαζόμαστε ε, μόνιμους ε, βοσκότοπους, βιοπικιλότητα, άνοιψη σπορά και πολλά ακόμα. Και αυτά θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε πώς οι στόχοι μας θα εξυπηρετηθούν από όλα αυτά έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τη δουλειά της. Ο κύριος Κούσμικ με εξέπληξε μεταφορά από το Ταμείο Συνοχής στη Γεωργία με μεγάλη χαρά. Γιατί ξέρετε πως το Ταμείο Συνοχής έχει πολλά κονδύλια και πάντοτε υπήρχε κάποιο είδους εξισορρόπηση, αλλά αν θέλετε να προτείνετε κάτι τέτοιο, καμία αντίρρηση. Τα Ταμεία Συνοχής να ε, αποδοθούν στην Γεωργία. Αλλά νομίζω ότι κάποιοι θα έχουν άλλη άποψη. Δίκη κατανομή πληρωμών. Πολύ το σχολιάσατε. και το έχουμε μπροστά μας στο έγγραφο. Τα στοιχεία στο, στο, στην πρώτη εκδοχή ήταν πιο συγκεκριμένα, αλλά ε, ήταν περισσότερο σκέψεις. Ε, τώρα για τη σταδιακή μείωση των πληρωμών, για την αναδιανομή, για τους μικρούς ε, γεωργούς, όλα αυτά θα πρέπει να τα αποφασίσουμε με τους συνομοθέτες. Δεν μπορούμε τώρα να βάλουμε νούμερα και εξαρτάται αν θα έχουμε υποχρεωτικά ή εθελοντικά ε, καθεστώτα και βεβαίως έχει να κάνει και με το πώς θα προχωρήσει η διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό. Θέλουμε να ακούσουμε και την άποψη των γεωργών. Νομίζω πως για την ευημερία των ζώων τα όσα είπατε είναι θετικά. Θα πρέπει τουλάχιστον να αναγνωρίσουμε πως υπάρχει τέτοιο θέμα και νομίζω ότι στο έγγραφό μας το αναγνωρίζουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε με κάποιες λύσεις που προτείνουμε και όλοι οι στόχοι, το λέω στην κυρία Ντελαχέ, θα είναι ευρωπαϊκοί και όλα τα σχέδια θα τα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε ελπίζω αυτό να σας δίνει, να σας καθησυχάζει. Δεν μιλάμε για επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ. Όχι, απλούστευση αυτής. Και συμφωνώ με τον κύριο Γιάρα. Βέβαια, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε να μην έχουμε νομοθετικό υπερθεματισμό, αλλά αυτό συμβαίνει και σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν στο μέλλον να σταθούμε πιο δραστήρια για να εξασφαλίσουμε πως όλη αυτή η απαραίτητη γραφειοκρατία που έχουμε επιβάλει στο Γιώργο είναι κάτι το οποίο θα διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά από ό,τι μέχρι σήμερα και θα είμαστε πιο δραστήριοι και εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων. Όταν δεν καταφέρνουμε τους στόχους μας, τότε ναι, έχουμε ένα εθνικό σύστημα κυρώσεων για το χρηματοδοτικό φάκελο. Ναι. Οπότε, αν μετά από κάποια χρόνια πετύχαμε τους στόχους μας και τις αποδόσεις, ναι. Αν όχι, τότε κάποια μέτρο, για παράδειγμα, όπως η αναστολή πληρωμών. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσουμε πως τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου ε, καταφέρνει αυτά τα οποία έχει θέσει ο στόχους και με τον τρόπο αυτό μόνο θα πιέσουμε όσους ε, ακολουθούν αυτή τη διαδικασία να κάνουν αυτά που πρέπει. Τώρα για τη μετανάστευση δεν είπα περισσότερη μετανάστευση, αλλά είπα πως η Γεωργία μπορεί στα πλαίσια των ε, επενδυτικών προγραμμάτων της, Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω της εξωτερικής, των εξωτερικών επενδύσεων που κάνουμε μέσω της ΕΤΕ να πετύχουμε τους στόχους μας. Μπορούμε να μοχλεύσουμε επίσης τα κονδύλια που έχουμε και με τη βοήθεια των φίλων ε, στην Αφρική και της ΕΤΕ να καταφέρουμε κάτι καλύτερο. Έχουμε εμπειρία και με γνώση που μπορούμε να μεταφέρουμε στις χώρες Αφρικανικής Υπήρου που κάνουμε σε κάποιες από αυτές αλλά όχι όσο θα έπρεπε, γιατί βεβαίως η παράδειγμα μετανάστευση θα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στο μέλλον αν δεν το αντιμετωπίσουμε σήμερα. Η Γεωργία έχει ένα ρόλο να παίξει και την έχουμε υποεκτιμήσει στο πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τις βασικές αιτίε που προκαλούν τη μετανάστευση. 60% της οικονομικής δραστηριότητας κάποιων αφρικανικών χωρών βασίζονται στη γεωργία. Και εδώ είναι οι νέοι, είναι οι γυναίκες, τους οποίους θα βοηθήσουμε με την προστιθήμενη αξία που έχει η γνώση μας. Θα μπορούν λοιπόν να καλλιεργήσουν τις δικές τους οδιές, να θρέψουν τις δικές τους γενιές και να ξεπεράσουν κάποια από τα προβλήματα που έχουν σε καθημερινό επίπεδο με τα κράτη-μέλη. Θα αντιμετωπίσει Συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε προβλήματα βρεθούν με την αγροτική ανάπτυξη και τα σχετικά προγράμματα με τα κράτη-μέλη, όχι με τις περιφέρειες. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Η μεταφορά κονδυλίων από τον ένα πυλώνα στον άλλο, ναι, γίνεται και σήμερα. Και δεν βλέπω να έχουμε κάποιε μεγάλε αλλαγέ εκεί, αλλά θα κοιτάξουμε του λόγου για του οποίου εσεί θέλετε να μεταφέρετε κονδύλια. Εμεί θα θέλαμε να γίνεται αν έχει ε, στόχο το περιβάλλον ή το κλίμα. Γιατί εκεί είναι η μεγάλη ευθύνη μας στην προστασία των πόρων για το μέλλον. Πολύ καλές ερωτήσεις μου κάνατε για την επικουρικότητα και για την εσωτερική αγορά. Ελπίζω να σας έχω καλύψει και ελπίζω να σας καθησύχασα. Για τη συγχρηματοδότηση νομίζω ότι ήταν ένα θέμα το οποίο θα δημιουργούσε πάρα, πολλά, πάρα πολλές αντιμαχίες είναι κομμάτι του εγγράφου προβληματισμού. Κάποια κράτη-μέλη το έθεσαν, αλλά αυτό θα πρέπει να το αποφασίσουν τα κράτη-μέλη τα ίδια. Στα πλαίσια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα πλαίσια της χρηματοδότηση μελλοντική ΚΑΠ. Και από τα στοιχεία που έχουμε στο τραπέζι θα δείτε ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα χάσουν. Και δεν νομίζω ότι εδώ υπάρχει περίπτωση να πετύχουμε μοφωνία. Αυτή τη στιγμή δημιουργούμε περισσότερα εργαλεία αγοράς για την αλυσίδα τροφής. Έχουμε το πρόγραμμα εργασίας για το 18, έχουμε το θέμα της διαφάνειας στην αγορά και των αθέμητων πρακτικών. Οπότε μπορούμε τώρα να ε, εξισορροπήσουμε την ισχύ του γεωργού σε σύγκριση με την ισχύ άλλων τμήματων της αλυσίδας διατροφής. Και πρέπει βεβαίως να εξετάσουμε ποιες προτάσεις μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε κρίσεις, να διαχειριστούμε κρίσεις σαν αυτές που περιγράψατε. Τώρα, για τον προπολογισμό είμαι μόνος. Και όταν έχει κάποιο το 38% του προπολογισμού, όλοι θέλουν να του φάνε κάτι. Εμεί, εν πάση περιπτώσει, στο τέλο τη ημέρα θα εξαρτηθούμε από το τι μπορούμε να κάνουμε για του άλλου επιτρόπου, αλλά η πρόταση αυτή είναι ένα κομμάτι τη εξίσωση. Τα κράτη-μέλη λαμβάνουν τι αποφάσει και το τι θα γίνει με τον προπολογισμό που θα λείψει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Brexit είναι θέμα κρατών μελών σε μεγάλο βαθμό. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και να, στο σημείο αυτό και να σας πω για τον κύριο Νταντά ότι... Πράγματι έγιναν συναντήσεις και στο, συζητήσεις και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι προφανές ότι η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας πρέπει να συνδυάσει τις προσπάθειές της και με τις υπόλοιπες γενικές διευθύνσεις και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό για να ξεπεράζουμε τις δυσκολίες και στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων. Στις σελίδες 17 και 18 περιγράφουμε τις λεπτομέρειες γύρω από αυτό. Τώρα θα πρέπει εμείς να δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτή την προσπάθεια και μπορούμε να βασιστούμε στη σωστή δουλειά η οποία έχει γίνει μέσω του Omnibus στα πλαίσια της διαχείρισης κρίσεων. Για την κυρία Μαγκίνες προφανώς αυτό το οποίο είπατε είναι πάρα πολύ σωστό. Ε, οι καινοτόμες πρακτικές θα πρέπει να υποστηριχθούν και ο νέος τρόπος λειτουργίας, το New Delivery System θα επιτρέψει να εφαρμοστούν αυτές οι προτάσεις ε, είναι ε, επιλογές που ανοίγονται έτσι ώστε να σεβαστούμε τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Θα δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να είναι και ευέλικτα και αυτή τη στιγμή εμείς θεωρήσουμε ότι έχουν πετύχει τους στόχους και μπορούν να εφαρμόσουν τους στόχους αυτούς σε τοπικό επίπεδο, τότε από εκεί και πέρα θα είμαστε διατεθειμένοι να ακούσουμε νέες προτάσεις και έτσι θα χρησιμοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε τις βέλτιστες πρακτικές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα μείνουμε στη λογική του ε, μία είναι η λύση που θα πρέπει να εφαρμοστεί για όλους. Τώρα, οι ορισμοί για τους γνήσιους γεωργούς Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες σε σχέση με τους ορισμούς. Νομίζω ότι καλό είναι να, τα κράτη-μέλη να μπουν στον κόπο να δώσουν εξηγήσεις σε σχέση με τον ορισμό του ενεργού α, ε, α, ε, ε, γεωργού. Δεν μιλάμε για επενδυτές, μιλάμε για γεωργούς και ιδιαίτερα νέους γεωργούς. Για το ανώτατα όρια και τα κάπινγκ, κύριε Φλάναγκαν, αναφέρθηκα ήδη. Αν είναι κάτι το υποχρεωτικό και το αποφασίσουν αυτό οι συνομοθέτες, τότε τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υπακούσουν. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το παρακολουθήσουμε αυτό και θα ελέγξουμε τα προγράμματα τα οποία θα υποβάλουν. Παρ' όλα αυτά είναι θέματα τα οποία μένει ακόμα να ειδωθούν. Εμείς έχουμε εντοπίσει κάποια θέματα σε σχέση με την, με την ισότητα, αν θέλετε, και τη δικαιοσύνη στην κατανομή των πιστώσεων. Φυσικά και θα πρέπει να στηρίξουμε και τους συνεταιρισμούς και τις οργανώσεις γενικότερα των παραγωγών, πρέπει να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα και εσείς αναφερθήκατε στο θέμα των, της δίκαιης κατανομής των πληρωμών. Ε, το θέμα είναι λοιπόν πως και εγώ και ο αρμόδιος υπουργός για θέματα ε, προϋπολογισμού ε, θα μπορέσουμε να ελέγξουμε λίγο το δημοσιονομικό βάρος. Το θέμα είναι να φτάσουν τα χρήματα στους γεωργούς και όχι στους επενδυτές. Δεν είναι αυτή η λογική οι γεωργοί θα πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα ωφελούνται από τα χρήματα τα οποία θα δόθηκαν. Υπάρχουν κάποια εθελοντικά προγράμματα τα οποία μπορεί να χρησιμεύσουν να εφαρμοστούν ευρύτερα στο μέλλον. Ε, λυπάμαι που ο κ. Φερνάντες δεν είναι πια εδώ σε σχέση με τα σχόλια ε, το, σε σχέση με αυτό το οποίο είπα ότι θα βοηθήσουμε τους μετανάστες και αυτό θα οδηγήσει στις αυτοκτονίες Γεωργών. Αυτά είναι πράγματα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να αποδεχθώ, είναι απαράδεκτα. Ε, δεν χρειάζομαι μαθήματα από τον κύριο Φερνάντες. Ξέρω τις πολύ δύσκολες προσωπικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρίσκονται οι Γεωργοί μερικές φορές χωρίς μικρόφωνο σχόλια από την αίθουσα με τα οποία συμφωνεί ο Επίτροπος Χόγκαν. Είπατε το πώς θα έχουμε στόχους και δείκτες οι οποίοι να είναι λειτουργικοί. Ακριβώς αυτό θα αποδείξει και την ε, αποτελεσματικότητα των στόχων, των μεθόδων που ακολουθούμε για να πετύχουμε τους στόχους. Έχουμε λοιπόν τους δείκτες επιδόσεων έτσι ώστε να συμφωνηθούν προγράμματα κοινά ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία να είναι άμεσα εφαρμόσιμα. Και έχουμε τα κριτήρια για να το πετύχουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται συνεχώς. Να πω επίσης ότι οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ έχουν συνεργαστεί επικοδομητικά μαζί μας. Για πρώτη φορά νομίζω ότι υπάρχει μια ευκαιρία να υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους εμπλεκομένους στην γεωργία και στο περιβάλλον. Ε, καταλαβαίνουν ότι και αυτοί που ασχολούνται με το περιβάλλον στις ΜΚΟ, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν τη γη είναι αυτοί οι οποίοι φροντίζουν το περιβάλλον, δηλαδή οι αγρότες. Αυτοί είναι οι θεματοφύλακες της ποιότητας του περιβάλλοντος και θα πρέπει φυσικά να πληρώνονται για να μπορούν ακριβώς να εξυπηρετούν τα οικοσυστήματα όπως πρέπει εξ ονόματος της κοινωνίας. Αυτό είναι η πρόκληση την οποία έχουμε σε δημοσιονομικό επίπεδο. Να πω τελικά κυρίες και κύριοι ότι πιστεύω ότι το θέμα της σύγκλησης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι ταυτόχρονα ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, αλλά νομίζω ότι προοδευτικά όπως είπε και ο κύριος Γιούνκερ προχωρούμε ε, σε μια πραγματική ε, ισορροπία στις πληρωμές, ισότητα στις πληρωμές ε, και νομίζω ότι εφόσον συμφωνούμε με το στόχο αυτό είναι ακριβώς ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε. Και αν μπορούμε να βρούμε περισσότερα χρήματα και μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς για διάφορες χώρες όπως η Βουλγαρία και άλλες χώρες, γιατί όχι, τότε θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο οι χώρες και οι καθαροί πληρωτές και οι καθαροί εισφορείς δηλαδή και οι υπόλοιπε χώρες πάρα πολύ δύσκολα θα αλλάξουν την πρακτική η οποία ακολουθείται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια πολιτική διαδικασία, θα πρέπει να γίνει μια πολιτική συζήτηση και θα δούμε ποια είναι η κατάληξη τη συζήτησης αυτής. Πάντως απαιτείται να υπάρχει μια σωστή χρηματοδότηση της κοινή αγροτικής πολιτικής έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό το οποίο και εσείς και εγώ επιθυμούμε μαζί. Ελπίζω να έχουμε μια καλή κοινή αγροτική πολιτική με μια Κύριε χρηματοδότηση. Κυρίες και κύριοι, ο Επίτροπος παρουσίασε την ανακοίνωσή του και βεβαίως αυτό έχει μια σημαντική πολιτική σημασία και βαρύτητα. Πρόκειται για ένα σημαντικό μήνυμα. Σας ευχαριστούμε που βρήκατε το χρόνο να έρθετε στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μαζί μας τις προτάσεις και τις θέσεις σας. Βεβαίως θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να διαβάσουμε προσεκτικά το κείμενό σας. Σίγουρα θα ακολουθήσουν πολλές ερωτήσεις, υπάρχουν αμφιβολίες, επιφυλάξεις, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η μελλοντική ισορροπία των δυνάμεων και δυναμική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως μέχρι το 2019, μέχρι τις εκλογές, θα πρέπει αυτή η νομοθετική πρόταση να προχωρήσει και συμφωνούμε μαζί σας ότι βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των μελών του Κοινοβουλίου, των κυβερνήσεων και ελπίζω να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό κλίμα για τη συζήτηση μέσα στην οποία θα εξελιχθεί η επεξεργασία αυτών των προτάσεων για την κοινή αγροτική πολιτική. Η χρηματοδότηση είναι κάτι πολύ σημαντικό και βεβαίως θα συναντήσουμε και τον αρμόδιο επίτροπο για θέματα προϋπολογισμού. Θα του θέσουμε ερωτήσεις. Ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό πριν τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές. Η επόμενη συνάντησή μας θα λάβει χώρα στις 3 την Δευτέρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες σας και ευχαριστώ και όλους τους εκπροσώπους της ΚΟΠΑ ΚΟΖΕΚΑ και όλους τους προσκεκλημένους μας σήμερα στην αίθουσα.